Colleagues, good afternoon. We've got... Καλό απόγευμα, κυρίε και κύριοι. Έχουμε μαζί μα του εισηγητέ για τα διάφορα προγράμματα ΔΕΔ. Έχουμε τον κύριο Μπάλα, τον κύριο Τελίτσκα και τον κύριο Μπρίνκχορστ. Θα μας μιλήσουν για 10 λεπτά και μετά θα δούμε. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Αύριο το πρωί έχουμε τους άλλους συντονιστέ. Τον κύριο Κόξ, την κυρία Πάης, τον κύριο Βαλέτε Ντιολιβέιρα και τον κύριο Σαβαρή και τον κύριο Βίντς. Και βεβαίως έχουμε και τον ε, ε, αντιπρόεδρο Κάλλας. Ε, αφού θα ακούσουμε λοιπόν όλους τους συντονιστές, θα έχουμε αυτό το ωραίο επιδόρπιο. Θα ακούσουμε τον Επίτροπο Κάλλας. Σχέδιο 17 είναι ο σιδηροδρομικός άξονας Παρίσι, Στρασβούργου, Τγκάρδη Βιέννη, Μπρατισλάβα. Κύριε Μπαλάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όταν ε, ε, σαν συντονιστές ε, μιλήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, το σημαντικό που προσπαθήσαμε να δείξουμε ήταν ακριβώς η προστιθέμενη αξία βάσει της προσπάθειας των κρατών μελών και της δικής μας βέβαια. Το PP17, Priority Project 17, πρόκειται για ένα ε, πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του σιδηροδρομικού ε, προγράμματος, καθώς επίσης ε, και της ανταγωνιστικότητας και της εσωτερικής αγοράς. Πολλά είναι τα στοιχεία της προστιθέμενης αξίας, κυρίως δε αυτό της διασύνδεσης κρατών μελών ε, επομένως, ε, μιλάμε για μια ανταγωνιστική υποδομή που καμία χώρα δεν μπορεί να στηρίξει από μόνη της. Ε, οι όμορες, οι γειτονικέ χώρες θα πρέπει να μπορέσουν να συζητούν μεταξύ τους και να καταλήγουν σε τέτοιου είδους προγράμματα. Το δεύτερο στοιχείο θέμενης αξίας είναι ότι ε, περνάμε στην διατροπικότητα, ξεπερνάμε δηλαδή τον σιδηροδρόμο από μόνο του. Έχουμε εσωτερικές πλωτές οδούς σε διασύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο, με τα αεροδρόμια, ε, με τους εξωτερικούς λιμένες κτλ. Τρίτο στοιχείο είναι η διασύνδεση ε, μεταξύ χωρών και δημιουργία ε, δικτύου σιδηροδρόμων. Και τελευταίο στοιχείο, αλλά όχι ελάσσονο σημασίας, ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει, είναι το, η, η επίτευξη μάλλον ε, συνέχειας, ε, έστω και αλλάζοντας χώρες, αλλά και αλλάζοντας κυβερνήσεις. Γιατί πρέπει να είναι μια γραμμή η οποία θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ ε, και ε, σημαντικών ε, πρωταγωνιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πιο ευάλωτων παικτών. Και μπορώ να σας δώσω ένα μακρύ κατάλογο πολιτικών και κυβερνητικών μελών Υπουργείων στις τέσσερις χώρες. Μπορώ να σας πω ότι τα κράτη-μέλη έχουν την βούληση να υλοποιήσουν το, κατά προτεραιότητα, το πρόγραμμα προτεραιότητας 17 διότι είναι επεπισμένα τα κράτη-μέλη ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για την Ευρώπη και για τα ίδια. Μέχρι τώρα 43% της γραμμής έχει ολοκληρωθεί και 44% εξακολουθεί να ε, κατασκευάζεται. Βεβαίως τα κράτη-μέλη συνειδητοποιούν ότι σε μια μεγάλη διακρατική γραμμή ε, τα διακυβεύματα είναι πολλά. Και βεβαίως ε, πρέπει να είναι σε θέση να ε, ολοκληρώσουν τις ε, διαδικασίες. Πρέπει να σας πω ότι και η Γαλλία ολοκληρώνει τη γραμμή ε, TGV, τρένου υψηλής ταχύτητας. Να σας πω όμως τα πράγματα αναχώρα. Στη Γαλλία έχουμε το TGV από το Παρίσι μέχρι το Ποτρεκούρ και το υπόλοιπο θα ξεκινήσει το 2012 με στόχο να έχει ολοκληρωθεί το 2016 που για τέτοιο, τέτοιο έργο υποδομής ε, είναι πολύ κοντινό. Έχουμε και το γαλλικό τμήμα λοιπόν το οποίο θα λειτουργεί πλήρως. Στην Αυστρία στο Σάνκτ Πέρτεν θα έχουμε έναν νέο σιδηροδρομικό σταθμό που θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο του 2000 ε, και τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε εγγένεια από το Σαντ Πέρτεν στη Βιέννη το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο. 8 Δεκεμβρίου του 2012 θα έχουμε τα εγγένεια. Και αυτό θα σημαίνει μείωση σημαντική του χρόνου ταξιδιού. Στη Γερμανία το πέρασμα του Ρήνου άνοιξε το Δεκέμβριο του 10, πριν από ένα χρόνο, ε, μία υπέροχη γέφυρα με διπλή γραμμή και επιτρέπει ταχύτητα της τάξης των 160 χιλιόμετρων οι εργασίες ε, των 61 χιλιόμετρων μεταξύ του Άξπορ και του ε, Μονάχου θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο. Ε, και αποτελεί το επιστέγασμα 13 χρόνων εργασίας. μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, τρέχοντο έτου δηλαδή, θα έχει τεθεί σε λειτουργία η γραμμή με τέσσερις ε, ε, τροχίες. Επίσης έχουν ξεκινήσει οι διασυνδέσεις ε, μεταξύ σιδηροδρόμου και αστικών μεταφορών. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην Γερμανία εν μέρη ε, στα τμήματα ε, τα συνοριακά της Γαλλίας και της Αυστρίας καθώς επίσης ε, και το, στο Appenweier. Και υπάρχει ένα τούνελ το οποίο ακόμα βρίσκεται υπό κατασκευή μεταξύ Μονάχου και Σάλτσμπουργκ θα ε, συνεχίσουν οι εργασίες. Αυτό που θέλουμε είναι να λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα αυτής της γραμμής. Δηλαδή, ο κεντρικός σταθμός στην πόλη της Τουσγκάρδης, ε, και οι διασυνδέσεις που θα φτάνουν μέχρι το σταθμό αυτό. Ένα δημοψήφισμα θα λάβει η χώρα σε μερικές μέρες από σήμερα, ε, τις 25 ε, Νοεμβρίου. Θα περιμένουμε λοιπόν την έκβαση του δημοψηφίσματος, θα περιμένουμε την ολοκλήρωση των πολιτικών διεργασιών και τέλος τις τεχνικές αποφάσεις. Η Σλοβακία παίζει ένα σημαντικό μέρος σε αυτό σε αυτή τη γραμμή γιατί στο τελευταίο, του κομμάτι, το τελευταίο της κομμάτι αυτή η γραμμή συνδέει δύο πρωτεύουσες, τη Βιέννη με την Πρατισλάβα. Υπάρχουν κάποιες περικοπές ε, στην ε, Πρατισλάβα. Πάντως νέες ναι, συζητήσεις έχουν ξεκινήσει στην Πρατισλάβα για το θέμα αυτό και για αυτό το, ε, αυτό το σχέδιο και Μέχρι το 2012 θα έχουμε το νέο μοντέλο ε, ε, συγκοινωνιών μεταξύ Βιέννας και Βρατισλάβα. Ε, και βεβαίως θέλουμε και διασύνδεση και με τα αεροδρόμια. Και βεβαίως για την Πρατισλάβα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό γιατί από μόνο του το αεροδρόμιο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί τόσο αποτελεσματικό από όσο όταν θα είναι διασυνδεδεμένο με τον σιδηρόδρομο. Επίσης ε, υπάρχουν πολλά αεροδρόμια ε, και πολλές εσωτερικές πιλωτές οδοί μεταξύ των οποίων ο Δούναβης και ο Ρήνος ε, και γίνεται προσπάθεια να διασυνδεθούν με την σιδηροδρομική τροχιά. Γίνονται επίσης ε, νέοι προγραμματισμοί όσον αφορά ε, την έκδοση εισιτηρίων, τη διακίνηση των επιβατών, έτσι ώστε ε, να είναι και καινοτόμα και πιο ελκυστικά. Επίσης νέες μορφές εισιτηρίων που θα συνδυάζουν το σιδηρόδρομο με το αεροδρόμιο και νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό και για τους ευρωβουλευτές που θέλουν να φτάσουν στο Στρασβούργο, γιατί θα υπάρχει μια καλή διασύνδεση μεταξύ ε, του σιδηροδρόμου και του αεροπλάνου, κυρίως ε, για τους βουλευτές ε, που προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα στην Αμβέρσα θα οργανωθούν οι γνωστές ημέρες ΔΕΔ, ε, με παράλληλα εργαστήρια και θα υπάρξει ένα εργαστήριο ακριβώς κατά αυτή την έννοια, διασύνδεση σιδηροδρόμου και αεροδρομίων και αεροπορικών μεταφορών. Πραγματικά προσδοκώ στη συμμετοχή σε αυτό το εργαστήριο γιατί πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, οι εκπρόσωποι των σιδηροδρόμων, εκπρόσωποι των αεροδρομίων, εταιρείε εμπλεκόμενες, ε, ε, κράτη πραγματικά θα μπορούν, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν έτσι ώστε ε, να ε, γίνει πιο απλό το ταξίδι ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης και αργότερα και πέρα από την Ευρώπη. Και βεβαίως όλα αυτά ε, προς διευκόλυνση των επιβατών που με πολύ απλό και εύκολο τρόπο θα μπορούν να πηγαίνουν από τον σιδηρόδρομο στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο και τούμπαλιν. Ε, αναφερόμαστε επίσης ε, σε διασύνδεση με λιμένες ε, που παραμένουν πολύ σημαντικοί σε, αυτήν, σε αυτόν τον άξονα του λεγόμενου αυτού που αποκαλούμε σήμερα Priority Project 17 και θέλουμε όλες οι διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το έτος 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπάλα. Έχω τρει ομιλητέ μέχρι στιγμή: Φέρμπερ, Κράμερ και Πίρκερ. Και την κυρία Λιχτεμπέργκερ. κύριο Φέρμπερ εκ μέρου του ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάλλας έναν από τους συντονιστές. Ε, πάρα πολύ ευρεία και εκτεταμένη η αναφορά που μας έκανε. Αυτό που έχει παρουσιάσει η Κομισιόν και έχουμε λάβει και εμείς, μας δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει μια παράλληλη διαδρομή, αν θέλετε, αν στη Βάλτε Βιτεμβέργη με το δημοψήφισμα δεν ε, δοθεί συνέχεια σε αυτό το έργο, στην εκτέλεση αυτού του έργου. Και η Στουτγάρδη 21 δεν είναι μόνο ένα σχέδιο που έχει να κάνει με το συνδεδρομικό σταθμό της Στουτγάρδης, αλλά με όλο το τμήμα του άξονα που φτάνει μέχρι τη Βαβαρία. Στον Γκάισλινγκε, που εκεί δεν μπορεί το τρένο να πάει πάνω από 100 χιλιόμετρα λόγω της κλίσης. και χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν δύο ε, μηχανές. Αυτό δεν είναι φυσικά ό,τι καλύτερο. Επίσης το τμήμα Μέσαρ, Μπρούκεν, Φραγκφούρτη ε, και τελικά Βιέννη θα αντικαταστεί στο τμήμα Στουτγάρδη Μόναχο. Από ό,τι φαίνεται, τι άποψη έχετε γιατί είμαι από το Χάψπουργκ και για το Αξπουργκ. Μιλήσατε για την περιοχή αυτή. Δεν θα ήθελα κάποια πράγματα να μείνουν στο περιθώριο. Ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστώ. Κύριο Σέρτουκα από την ομάδα των Σοσιαλιστών για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλλας και εγώ από την πλευρά μου ε, θέλω να σας ε, ευχαριστήσω για την εντυπωσιακή περιγραφή της κατάστασης για τον διάδρομο αυτό. Είπατε ότι έχει ολοκληρωθεί το 47% και το 44% ε, από ό,τι κατάλαβα έχει δρομολογηθεί για όλο το τμήμα. Έχω κάποιες ερωτήσεις, θα επικεντρωθώ στα σημαντικότερα ερωτήματα και ιδίως στο κομμάτι μεταξύ ε, Στρασβούργο Απλμπάι, Μιλήσατε για το Κέλ Απλμπάι, αλλά Έχουν ηλεκτροδοτηθεί και δύο γραμμές από ό,τι κατάλαβα, αλλά δεν έχω καταλάβει κάποια πράγματα. Πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα σε σχέση με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο δηλαδή. Τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς για να στηρίξουμε εάν πρέπει να στηρίξουμε αυτό το έργο. Εγώ είμαι επίσης από τη Βαβαρία και θα ήθελα να δω τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο τμήμα τώρα, Μόναχο Μόναχο-Σάλτσπουργκ. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός διάδρομος αυτός, γιατί συνδέει το Μόναχο με ένα τρίγωνο εκεί και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι μελέτες. Το θετικό σε όλα αυτά είναι ότι το Δεκέμβριο του 2010 αποφασίστηκε η διεύνηση ενός τμήματος που όμως δεν λύνει τα προβλήματα που έχουμε στη Γερμανία με τη συμφόρηση, με τις εμπορευματικές μεταφορές, μεταφορές επιβατών, τεράστια κυκλοφορία και ροή. Πώς ε, προχωρούν διαπραγματεύσεις με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών. Μίλησατε επίσης ε, για τη σειρά καράστα. Δύο έργα προτεραιότητας είναι το PB7 και το 24 Χθε όμως ε, ακούσαμε από το γερμανικό τύπο ότι αυτό το συνδεδρομικό τούνελ θα γίνει εκεί που έχει προβλεφθεί και εξέφρασαν την άποψή τους και οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι. Εσείς τι νομίζετε, θα δώσει όμως για κυβέρνηση χρηματοδότηση. Τι θα συμβεί. Ευχαριστώ κύριο Σκράμερ. τρία λεπτά τώρα, Μίχαηλ, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κράμερ. Ίσως αυτές να είναι και οι τελευταίες πληροφορίες από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών που μάλλον φαίνεται να γνωρίζει καλά τα πράγματα που έρχεται και από την Βαβαρία. Τι κάνουμε τώρα. Εσείς είπατε ότι το 40% είναι έτοιμο και λέτε All are willing to do that. Ε, όλοι δηλαδή είναι πρόθυμοι να το κάνουν αυτό. Ξέρετε όμως ότι ναι μεν έχουν υπογραφεί κάποιες συμβάσεις, αλλά δεν ε, αρκεί υπογραφή, δεν αποτελεί απαραίτητη εγγύηση για το ότι θα ολοκληρωθεί. Στη Γερμανία λέμε ότι θέλουμε 7 δις για να αλλάξουν ε, κάποιες υποδομές, αλλά δεν υπάρχουν. Αυτή η λύση που προτείνει ο κ. Φέρμπερ ε, πρέπει να τη συζητήσουμε, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι που έχει γίνει κατά το ίμιση μεταξύ Νιρεμβέργης Μονάχου Βίρτσμπουργκ. Είναι έτοιμα αυτά τα κομμάτια. Δεν ήθελα να μου πείτε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, ακόμη κι αν δεν είναι ικανοποιημένος ο Σναβαλόμος, τι κάνουμε. Γιατί στο Τουτγάρδη μιλήσατε για αυτό το πρόβλημα, το σχέδιο Τουτγάρδη 21, ο συνδεδομικός σταθμός, ο κεντρικός, δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι ε, έχει γίνει σε άλλα κρατημέλη. και για τον Γκάι Σιγκεστάιγκε. Φυσικά και δεν είναι πρακτικό. Αλλά η άλλη πρόταση, ούτε και αυτή είναι πιο πρακτική. Έχουμε τρία δις σε μια διαδρομή που τελικά δεν πρόκειται να λειτουργήσει από ό,τι φαίνεται. Όχι, δεν είπα ότι είπατε κάποια ανοησία, αλλά τέλος πάντων, εγώ επειδή έχω το λόγο θέλω να με πρέπει να ολοκληρώσω. Πώς πρέπει να προχωρήσουμε, αυτό είναι το θέμα. Η νομοθεσία που προβλέπετε, ότι οι σταθμοί ε, ή τυπώγεται όχι, ε, πρέπει να πληρούν κάποια πρότυπα, πρέπει να πληρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όλα αυτά έχουν εγκριθεί. Τα έχει υπογράψει η γερμανική δημοκρατία. Όμως, η Στουτγάρδη δεν σέβεται αυτά τα πρώτα αυτούς κανόνες. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψή σας και τι προβλέπετε πάνω απ' όλα, τι προβλέπετε ε, σε σχέση και με το δημοψήφισμα που θα γίνει στη Στουτγκάρδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, να επενθυμίσω σε όλους ε, ότι ό,τι σχολείτε να κάνετε, ακόμη και αν θέλετε να προσβάλλετε κάποιον, να απευθύνεστε προ το Πρόεδρο, παρακαλώ. Κύριο Σπίρκερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω και το, τον συζητητέ και του συντονιστέ. Έχω τρει ερωτήσει. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά αυτό το σημείο, το, σημείο, το ανοιχτό μεταξύ Φράι Λάσεν και Σάλτσμπουργκ. πρέπει να γίνει ε, αυτή η γέφυρα πάνω από το Σάλαχ. Ε, η Αυστρία έχει κάνει τα απαραίτητα, αλλά η γέφυρα δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί. Για ποιο λόγο. Πότε περιμένουμε να ξεκινήσει η κατασκευή. Πότε θα έχει ολοκληρωθεί λοιπόν και σε ό,τι αφορά την διασύνδεση με τον αερολιμένο, με το αεροδρόμιο. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και με τη σύνδεση με την Αντριατική και μέχρι την ε, Μπρατισλάβα. Στην έκθεσή σας βλέπω ότι πρόκειται να υπάρξουν και άλλες συζητήσεις λόγω της οικονομικής αξιολόγησης της κατάστασης και ίσως τα έργα τροποποιηθούν Άρα, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Τα δύο αεροδρόμια της Μπρατισλάβα με τη Βιέννη πότε θα διασυνδεθούν και αν υπάρχει καθυστέρηση που οφείλεται αυτή. Το επόμενο ερώτημά μου. Διατροπικότητα. Αναφέρατε τη λέξη αυτή και πραγματικά εδώ στην ε, Επιτροπή μας και στην, ε, στον τομέα των μεταφορών μας ενδιαφέρει πάρα πολύ Έχουμε το συνδυασμό ε, των οδικών, ισοδρομικών, θαλάσσιων μεταφορών. Τι προκαταρκτικό έργο θα αναλυφθεί στο άμεσο μέλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί βέλτιστα, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Κύριε Λιχτεμπέργκερ, κάποια από τα ερωτήματά μου έχουν ήδη τεθεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάντως ε, που συμπεριλάβατε αυτό το τρίγωνο, ε, το τρίγωνο της, ε, το χημικό, ε, που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό έργο. Και έτσι έχουμε εδώ ένα σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει βέβαια και με τη μεταφορά επιβατών στην περιοχή αυτή. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα. Δύο ρωτώ με, επειδή ταξιδεύω πάντα με το τρένο για το Στρασβούργο. Τι θα γίνει μετά από τη γέφυρα με το ΚΕΛ, δεν έχω καταλάβει ακριβώς ε, τι γίνεται. Και το τρίτο, σε σχέση με το κομμάτι Βιέννη Μπρατισλάβα. Δεν είναι σαφής η προτεραιότητα από ό,τι φαίνεται μεταξύ των εταίρων, γιατί φαίνεται να υπάρχουν ε, διαφορετικά μηνύματα ε, στην ε, Αυστρία ή στη Σλοβακία. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει. Το θέμα είναι να γίνει μια γρήγορη διασύνδεση μεταξύ των δύο αυτών πόλεων. Είναι και ο καλύτερος ε, διάδρομος. Οι βελτιώσεις έχουν ήδη επιφέρει ε, βελτιώσεις της μεταφάσης επιβατών και εμπορευμάτων. Γίνονται δηλαδή κάποια πράγματα, βλέπουμε καρπούς, παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η γραμμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε, κύριε Συντονιστά. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο ενώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής σας, ήμουνα όμως παλιότερα, 10 χρόνια μέλος. Και έτσι θεωρώ ότι έχω το δικαίωμα να ρωτήσω τα εξή. εσείς λέγαμε τόσα χρόνια. Όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε συστήσει τόσο καιρό. Έχουμε συστήσει τη χρηματοδότηση. Έχουμε συστήσει όλα τα προβλήματα με μεγάλη σοβαρότητα όλα αυτά τα χρόνια. Εσείς εκπροσωπούσατε εκ μέρους της Βάδης Φιτεμβέργη την σοβαρότητα, τα, τη σοβαρότητα Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι όσα λέγαμε μέχρι τώρα, όσα κάναμε, όσα απαιτούσαμε, σε σχέση με τον στερεονομικό άξονα Παρίσι Τρασβούρου, Τικάρδη Βιέννη Βρατισλάβα, φαίνεται ότι ήταν όλα ανοησίε. Παρακαλώ λοιπόν να μα πείτε ξεκάθαρα. Εάν όλα αυτά για τα οποία έχουμε τόσο σκληρά αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια είναι ρεαλιστική πραγματικότητα, είναι μια καλή βάση ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. τρία δευτερόλεπτα. είχατε πει ότι πρέπει να περάσει από το Σφέχαρτ μετά προς τα νότια η γραμμή αυτή Βρατισλάβας Βιέννης. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει. Mr. Ballas, was 18, but I grant you. ήταν ο λοιπάς κύριε Μπάλλας. Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Μία συζήτηση με τον Υπουργό όμω. Είναι απαραίτητο πιστεύω. Και έχω ένα κατάλογο ερωτήσεων. Σε ένα βαθμό τις επιβεβαιώσατε. Θέλετε κι εσείς να έρθετε εδώ κύριε Μπάλας. Ίσως να προσθέσω και άλλες ερωτήσεις αν έχετε κάποια εκκρεμότητα στον κατάλογο μου. Εν περιπτώσει θα ήθελα να περιοριστώ μόνο στην εντολή μου για το σχέδιο προτεραιότητας 17 και σε αυτό απαντώ μόνο. Έχετε προσθέσει βέβαια νέες πτυχές, νέες πτυχές, νέες ερωτήσεις με τις παρατηρήσεις σας. Για ορισμένα ζητήματα δεν μπορώ να πω ότι είχα την ευκαιρία να συζητήσω προσωπικά με τον Υπουργό. Πάντως είμαι διατεθειμένος ανά πάσα στιγμή να μεταβώ είτε στο Βερολίνο είτε σε οποιαδήποτε άλλη γερμανική πόλη. Τελευταία φορά είχαμε την ευκαιρία να τεθούμε στο Στρασβούργο. Ήταν μια καλή ιδέα εκτός των συνόρων, συζήτηση, καλή συζήτηση, φιλική συζήτηση, αλλά και στο Βερολίνο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν τόντι ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Γερμανίας. Τις αρμοδιότητες από την άλλη των κρατηδίων Έτσι και η Επιτροπή ή ένας ε, μεμονωμένος συντονιστής σίγουρα δεν μπορεί να κρίνει τα θέματα αυτά. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι μια, να σας δώσω μια εικόνα της κατάστασης όπως την καταγράφω εγώ. Αλλά και εγώ έχω τους προβληματισμούς μου και τα ερωτηματικά μου προς τα κρατη Και πρώτα απ' όλα προς τον Υπουργό των Μεταφορών της Γερμανίας θα έστρεφα τις ερωτήσεις μου. Γιατί δεν συνεχίστηκαν οι εργασίες. Δεν ξέρω να σας πω εγώ προσωπικώς. Είχε προβλεφθεί αρχικά ότι θα ήταν πρώτα έτοιμη αυτή η πολύ ωραία γέφυρα στο Κιλ. Δεκαετίες πέρασαν Έγιναν μεγάλες εκδηλώσεις, πανηγυρισμοί, είχαμε δύο λωρίδες, ταχύτητα 160 χιλιόμετρων και μαζί με τον κύριο Ράμσα τα εορτάσαμε όλα αυτά και μετά από τους εορτασμούς σταμάτησαν οι εργασίες, δεν προχώρησαν περαιτέρω. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και αλλού. τον Geisling και Έτσι λοιπόν, δεν θα επαναλάβω όλα αυτά τα ερωτήματα. Θα ήθελα ωστόσο να πω ότι εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από διάφορες πλευρές και από τους τουριστές βεβαίως θεωρώ ότι πρέπει να τίθενται διαρκώς τα ερωτήματα αυτά. δεν υπάρχει γραμμή που να μην είναι σημαντική, εν προκειμένου. Αν δεν αναπτυχθεί ολόκληρη γραμμή, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έτσι. Υπάρχουν ε, σημεία της γραμμής που χάνεται η ταχύτητα στην ε, Βαβαρία, όπως στο τριγώνο του Χέμι παραδείγματι. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πρέπει να δεχθούμε ότι έχει αρμοδιότητα το κράτος, έχει αρμοδιότητα το κράτος μέλος, ε, ο καθένας έχει τις αρμοδιότητές του δηλαδή και πρέπει να συνδυαστούν αυτές. Εγώ τώρα ως συντονιστής επισκέφθην την ε, Στουτχάρδη και όταν είχα πάει εκεί το 2005 πρώτη φορά, η πρώτη μου ερώτηση ήταν τι εναλλακτικέ έχουν σχέση με το σχέδιο αυτό. Η απάντηση ήταν δεν υπάρχει εναλλακτική. Ουδέμια. Αυτό σε πολιτική ορολογία σημαίνει ότι έχει ληφθεί η απόφαση. Είναι τελεσμένη και πρέπει να τηρηθεί. Και δεν υπάρχουν εναλλακτικέ, μου λεγόταν. Όμω εναλλακτικέ υπάρχουν πάντοτε. Μια νέα πολιτική κατάσταση επιτρέπει και λόγω των διαφόρων ε, διαμαρτυριών και αντιδράσεων που ανεπτύχθησαν στη Σουτχάρδη να αναζητηθούν άλλες εναλλακτικές. Και νομίζω ότι για την αλλαγή δεν χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο. Τα, τα γερμανικά δεν είναι μητρική μου γλώσσα. Είναι μια γλώσσα που αγαπώ πολύ και μιλάω πολύ όταν έχω την ευκαιρία. Αλλά όταν μιλούμε για άσκηση του δικαιώματο της καταγγελίας συμβατικών υποχρεώσεων για το συντηροδρομικό σχέδιο στο ΤΧΑΡΤΗ 21, είναι σαφές νομίζω, έστω και χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο να δώσει κανείς την νομική ερμηνεία αυτής της φράσεως, της νομικής φράσεως που είναι τόσο περίπλοκη. Είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει κανείς να περιμένει πρώτα απ' όλα το αποτέλεσμα αυτής ε, της μορφής δημοψηφίσματος, του του. και στη συνέχεια πολιτική ερμηνεία της έκβασης του δημοψηφίσματος και την για να δούμε και την αντίδραση της τοπικής κυβέρνησης του κρατηδίου για να ακολουθήσει μετά η επόμενη φάση της τεχνικής προσαρμογής της πολιτικής αποφάσεως. Περαιτέρω ζήτημα αυτό, πώς δηλαδή θα υλοποιηθεί, πώς θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό, αυτή η απόφαση, όποια απόφαση Άρα θα πρέπει να επανέλθει φαντάζομαι σε ε, συγκεκριμένη χρονική στιγμή με το θέμα αυτό και πάλι για να σας δώσω τις περαιτέρω πληροφορίες για την υπόθεση αυτή. Για το αν υπάρχουν εναλλακτικέ οδοί, η απάντηση που θα να σα δώσω είναι όχι με βάση τη δική μου εντολή. Η δική μου εντολή μιλάει για Παρίσι ή Μπρατισλάβα. Άλλη εναλλακτική δεν αφήνει. Στη ζωή εναλλακτικέ υπάρχουν πάντα. Διαφορετικέ επιλογέ υπάρχουν πάντα. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα δίκτυο το οποίο επιτρέπει βέβαια πάντα την αναζήτηση και εξέβρεση διαφορετικών επιλογών. Ένα λεπτό ακόμη αν μου επιτρέπετε. Μεταφορές φορτίων και τρίγωνο χέμι θα έλεγα επιτρέπουν μια διαφορετική προσέγγιση και θα ήθελα να πω ότι ο, η διασύνδεση των δύο αεροδρομίων έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα για την Πρατισλάβα και έχουμε προσπαθήσει δεδομένου ότι η διασύνδεση με το Σφέχαρτ και το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα φαινόταν δύσκολη υπόθεση τότε. Ε, μεταξύ βεβαίω έχει προχωρήσει η τεχνολογία, έχουν προχωρήσει και οι Υπουργοί Τεχνολογία της, ε, Μεταφορών της ε, Σλοβακίας, έχουν αλλάξει τα πράγματα δηλαδή και άρα μπορεί μετά τις εκλογές του Μαρτίου μια νέα ε, κυβέρνηση να δώσει διαφορετικές απαντήσεις οπότε και εγώ είμαι έτοιμος να μεταβώ εκεί ώστε να συζητήσω νέες λύσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλας. Περνάμε τώρα στο πρόγραμμα προτεραιότητας 27. Δηλαδή η Βαρσοβία, Κάουνας, Ρίγα, Ταλίν, Χελσίνκι. Ο κύριος Τελίτσκα έχει το λόγο. Παρακαλώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι μέλη του Κοινοβουλίου. Πρώτη φορά συμμετέχω σε συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τώρα καταλαβαίνω ότι μεταξύ ημών βρίσκονται και άνθρωποι οι οποίοι για χρόνια ασχολούνται με τα προγράμματα αυτά. Ε, αυτό σημαίνει ότι πολλά ενδιαφέροντα μπορεί κανείς να κάνει συνεργαζόμενος με το Κοινοβούλιο. Ε, και βεβαίως καταλαβαίνετε κι εσείς ότι και πρόοδοι έχουν γίνει, αλλά εξακολουθούμε να αντιμετωπίσουμε και κάποια ε, προβλήματα. Εγώ λέω πάντα έχει γίνει πρόοδος, αλλά υπάρχουν και κάποιες οπισθοδρομήσεις. Όμως, σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, μπορώ να πω ότι αυτή τη φορά παρά την δυσχερή οικονομική κατάσταση, κυρίως στις χώρες της Βαλτικής, ε, πρέπει να ομολογήσω ότι ε, υπήρξαν κάποιες ε, καλές αλλαγές και υπήρξε πρόοδος. Να υπενθυμίσω το, το πρόγραμμα Rail Baltica είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ε, έχει στόχο να ε, ενσωματώσει τις ε, νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες της Βαλτικής αλλά και την Πολωνία. Εδώ μιλάμε λοιπόν για χώρες οι οποίες έχουν πολλά συστήματα μονής τροχιάς και διπλής τροχιάς, ηλεκτροδοτούμενο και μη. Επομένως καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μείγμα ε, το οποίο δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει κανείς. Από την άλλη πλευρά και τα οικονομικά συμφέροντα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν οπωσδήποτε και κάποια ε, εκπεφρασμένα συμφέροντα τα οποία προσπαθούν ε, να βρουν το δρόμο τους στο σχέδιο αυτό. Ε, και ε, βεβαίως έχουμε αντιμετωπίσει και τον ανταγωνισμό ε, σε όρους γιατί οι γείτονές μας και όχι εμείς και καλύτερα εμείς και όχι οι γείτονές μας. Ε, υπενθυμίζω ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση με μεγάλη οικονομική ύφεση και βεβαίω αντιμετωπίζουμε και προβλήματα αλλαγή πολιτική ηγεσία. το ανέφερε αυτό και ο κύριο Μπάλλα προηγουμένω. Έστω όμω και με όλε αυτέ τι δυσκολίε έχει υπάρξει κάποια πρόεδρο. Θα είμαι λίγο πιο σαφή τώρα. Την προηγούμενη φορά που με καλέσατε εδώ και σας είπα ότι είχαμε κάνει αρκετή πρόοδο στην Εστονία, ήταν σαφές. Α, τώρα μπορώ να σας πω ότι πήγαμε παραπέρα, ότι μάλλον έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τη δουλειά στην Εστονία. Ε, μιλάμε τώρα για ταχύτητες 250 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα ε, στην ε, ολοκλήρωση ενός πράγματος που πριν από μερικά χρόνια ήταν στη σφαίρα της ουτοπίας και με τον τρόπο αυτό ε, να ενσωματωθεί η χώρα αυτή στο υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως ε, πρέπει να προχωρούμε προσεκτικά με σύνεση βήμα-βήμα έτσι ώστε τα, τα ε, σχέδια που κάνουμε να είναι σε θέση να επιβιώσουν οικονομικά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν στην, στην Εστονία και μάλιστα οι Εστονοί κατάφεραν να βάλουν και στην άκρη να αποταμιεύσουν ε, κάποια χρήματα. Έγινε λοιπόν πάρα πολύ σωστή η δαπάνη των ε, ε, χρημάτων. Λετωνία. Η Λετωνία είναι μια χώρα που όπως ίσως θυμάστε ζήτησε μια στάση του προγράμματος λόγω οικονομικών δυσχεριών. Είναι μια χώρα η οποία σε σύγκριση με τις άλλες χώρες ε, έχει μια αρκετά καλή σιδηροδρομική κατάσταση, αρκετά καλό σιδηροδρομικό ε, ε, δίκτυο, αλλά, αλλά στην παρούσα οικονομική κατάσταση το να φτάσουν στο επίπεδο του Rail Baltica θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Η, κυβέρνηση τον Απρίλιο πάντως αποφάσισε να ξαναρχίσει τις εργασίες και ε, να χρησιμοποιήσει 21,5 εκατομμύρια ε, από ίδια χρηματοδότηση. Εάν θέλετε μια αξιολόγηση από τη δικιά μου, μια εκτίμηση από τη δικιά μου πλευρά, ε, θα μπορούσα να σας πω ότι ναι, εάν εξακολουθεί η εφαρμογή των συμφωνηθέντων και εάν η κυβέρνηση επιβεβαιώσει αυτά που έχει αναφέρει, ναι, μπορούμε να μείνουμε στις οικονομικές προοπτικές. Εστονία. Ε, πριν από μερικούς μήνες είδαμε το άνοιγμα των πρώτων 106 χιλιόμετρων Ε, το νότιο τμήμα της Λιθουανίας, το νότιο τμήμα της Λιθουανίας ε, μέχρι τα σύνορα σχεδόν με την Πολωνία. Ε, με στόχο βέβαια να φτάσουμε στο Κάουνας. Έγινε μία επανεκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση και αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές ε, και να γίνει προσπάθεια μείωσης του προβλεπόμενου κόστους. Ε, επομένως, ε, συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής. Η άλλη απόφαση η οποία ελήφθη, που είναι επίσης σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, η λιθωνική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο ε, θεώρησαν το Rail Baltica ε, σαν ε, εθνική στρατηγική σχέδιο έτσι ώστε να ξεκινήσει και το θέμα της δίμευσης της περιουσίας, της απαλωτρίωσης μάλλον, που αποτέλεσε πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Τρίτη σημαντική απόφαση ή εξέλιξη στην ε, Λιθουανία ήταν ε, μία απόφαση που μπορεί ε, να είναι σημαντική, αλλά παρόλα αυτά έχει το, την αξία της αναγνώρισης του τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή, μία απόφαση της κυβέρνησης να χτίσει στο Κάουνις ένα κέντρο επιμελητίας Και γιατί είπα ότι μπορεί κανείς να γελάσει με αυτό. Είχαμε δύο σημεία, ε, το Μποντ και το Καρμέλεβα, που έριζαν για αυτό το κέντρο ευμιλητίας, αλλά τώρα ελήφθη η απόφαση ε, και επομένως με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει ε, το πρόγραμμα Rail Baltica να χρησιμοποιήσει ε, και την επιμελητία, Δηλαδή θα έχει και τη νέα υποδομή των σιδηροδρόμων αλλά και το κέντρο της επιμελητείας που δεν ήταν σαφές πριν. Στην Πολωνία τώρα. Είναι η μόνη χώρα, όπως γνωρίζετε ίσως, που αποφάσισε στα πλαίσια αυτού του σχεδίου να χρησιμοποιήσει το Ταμείο Συνοχής και όχι το ΔΕΤ Για περιβαλλοντικούς λόγους ελήφθη η τελική απόφαση να ε, ε, οικοδομηθεί νέα υποδομή κοντά στα σύνορα με την Λιθανία. Και βεβαίως ε, είναι μια ορθή απόφαση γιατί πρόκειται για μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή. η απόφαση αυτή οπωσδήποτε θα έχει επιπτώσεις στις ε, ε, μελλοντικές οικονομικές προοπτικές, αλλά πάντως ε, το σκεπτικό αυτής της απόφασης ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό που θέλουμε εμείς να διασφαλίσουμε είναι ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα και στις επόμενες μεσονομικές προοπτικές. Αυτά λοιπόν συνέβησαν με λίγα λόγια, αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, αλλά υπάρχει και μία μεγάλη ε, εξέλιξη που λόγω του ότι ε, πολύ νωρίς το Νοέμβριο έπρεπε να τυπωθεί η έκθεση, δεν ε, την λαμβάνει υπόψη. Η υπήρξε μία συνάντηση των εκπροσώπων των χωρών της Βαλτικής με τον Επίτροπο Κάλλας ε, και ε, εκπονήθηκε μία κοινή δήλωση ε, αυτό συμπίπτει με την ε, ε, δημοσίευση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας που χρηματοδοτήθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την, της χώρας της Βαλτικής. Πρέπει να σας πω ότι παλιότερα είχαμε τρεις ξεχωριστές μελέτες, τώρα έχουμε μία μονάχα. Και τα συμπεράσματα της ε, ε, της μελέτης αυτής ε, είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Βλέπουμε ότι είναι πιο, έχει μεγαλύτερο εύρος και καταλήγει στο ότι συμφωνούν όλοι σε διπλή ηλεκτροδοτούμενη ευθεία γραμμή από το Τάλιν ε, μέχρι τα σύνορα με την Πολωνία. Ε, και η, σύμφωνα με την μελέτη η λύση είναι βιώσιμη οικονομικά, μπορεί να αποτελέσει μία πάρα πολύ σημαντική επένδυση που θα ξεπεράσει τα 3,6 δις ε, ευρώ, αλλά θέλω να είμαστε προσεκτικοί με, το, με τα αριθμητικά στοιχεία. Μπορεί να είναι και λιγότερο, μπορεί να φτάσει και στα 6 δις. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα, προ, ένα σχέδιο το οποίο ε, θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα για σιδηροδρομικές ε, διασυνδέσεις μεγάλης ταχύτητας και θα φτάσουμε από να, να χρειαζόμαστε 8 λεπτά από το Ταλίν μέχρι τις, ε, τα σύνορα με την Πολωνία. Και επομένως την ερώτηση αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί η οικοδόμηση του Rail Baltica, εκεί η απάντηση σαφώς είναι ναι ε, ε, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει με το 2030 και θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε προσεκτικά και βήμα προς βήμα. Όσον αφορά τώρα τις πολιτικές ηγεσίε. είχαμε την ε, ε, πρωτοβουλία του Επιτρόπου ε, να συμπεριλάβει το Rail Baltica στις συζητήσεις και κατέστη φέσο ότι είναι για όλους ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και βεβαίως εξίσου σημαντική και η άλλη διάσταση Βαλτικής Αδριατικής. Επομένως, οι, ε, οι πολιτικές ηγεσίες των χωρών της Βαλτικής αποφάσισαν, πήραν αποφάσεις οι οποίες πριν από μερικά χρόνια ε, θα ήταν πραγματικά της σφαίρας της φαντασίας. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ε, σημείο, είναι μια καλή εξέλιξη. Ε, έχει προσκληθεί και η Πολωνία να συμμετάσχει σε αυτήν ε, την ομάδα ε, σκέψης των και βεβαίως έχει κληθεί και για το επόμενο κομμάτι και η Ιταλία και η Τσεχική Δημοκρατία, αλλά αυτό είναι μια άλλη διάσταση. Θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε κάνοντας κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι φυσικά ε, εξακολουθεί να είναι ένα πολύ δύσκολο ε, σχέδιο, αλλά ε, όπως καταδεικνύεται και από σχετικές μελέτες, είναι ένα σχέδιο με μεγάλη στρατηγική σημασία. Είναι, και είναι σημαντικό ότι υπάρχει η πολιτική βούληση και η φιλοδοξία έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το σχέδιο αυτό το πρόγραμμα που προτείνει ο Αντιπρόεδρος Κάλλας με βρίσκει ε, σύμφωνο και δεν είμαι, ξέρετε, πολύ εύκολος ε, στο να πείθομαι. Πάντως ε, είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, μια ενδιαφέρουσα αντίληψη του του πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε προβλήματα, το πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας σε γενόμενη όλο και πιο ανταγωνιστική στο μέλλον. Ε, φυσικά υπάρχουν ακόμα προβλήματα, προβλήματα τα οποία συνδέονται ε, με εκπεφρασμένα συμφέροντα και με άλλες δυσκολίες, αλλά είναι αντιμετωπίσιμα όλα αυτά. Τελευταία ε, παρατήρηση θα πρέπει να εφαρμοστούν όλες οι αποφάσεις. Δεύτερον, θα πρέπει να αρχίσουμε τον σχεδιασμό ε, του, της νέας διασύνδεσης ε, Βαλτικής ε, Αδριατικής. Τρίτον, να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο το ζήτημα της μεταφοράς επιβατών και να ξεκαθαρίσουμε το κομμάτι αυτό της Πολωνίας ε, που θα εμπέσει στις ε, ε, μελλοντικές, στις επόμενες χρηματοδοτικές προοπτικές και νομίζω ότι τελευταίο σημείο και πολύ σημαντικό ε, είναι ακριβώς να τονίσουμε το πόσο σημαντικό είναι πλέον που υπάρχει πολιτική βούληση, που οι ηγεσίε των τριών χωρών συνεργάζονται με τον Αντιπρόεδρο Κάλλας. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζασάντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Στονστό, δεν θα πρέπει να χρειάζεται πειθό κανείς για να φτιάξει διαδρόμους από βορρά προς νότο. Αυτό θα έπρεπε να εσύ και για την ε, Βαλτική και για το Rail Baltica δηλαδή. Πρόκειται για διαδρόμους οι οποίοι είναι απαραίτητοι και θα βοηθήσουν πάρα πολύ την κυκλοφορία στις, ε, και τις μεταφορές στις περιοχές αυτές. Για το σχέδιο προτεραιότητας λοιπόν το 27 του Rail Baltica σημειώνω βεβαίως ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Πολωνία όπως και για άλλες χώρες και των ε, ανατολικών βεβαίως κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν μέχρι στιγμής πολύ περιορισμένες δυνατότητες συνδροδρομικών μεταφορών, είτε φορτίου είτε επιβατών. Το υπόβαθρο το γνωρίζουμε βεβαίως αυτές τις υπόθεση, δηλαδή ήταν περιορισμένες και μόνο κατευθυντικές αυτές οι μεταφορές ε, στην παλαιά Σοβιετική Ένωση και τα παλιά Σοβιετικά κράτη. Έτσι λοιπόν δεν αναπτύχθηκαν ε, δίκτυα και αντίστοιχα και κοινότητες ε, που να βρίσκονται κοντά στην Δυτική Ευρώπη. Τώρα έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση και έτσι και εμείς ε, της Ανατολικής Ευρώπης ερχόμαστε πιο κοντά στη Δυτική. Όμως το σχέδιο αυτό έχει και μεγάλη οικονομική σημασία. Μεγάλη οικονομική σημασία ιδιαίτερος στις δεινές περιόδους που ζούμε Και γι' αυτό θα ήθελα προς το συντονιστή να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Η εφαρμογή του Rail Baltica και ο τρόπος που επηρεάζει τα κράτη-μέλη στην ε, περιοχή της Βαλτικής. Θα ήθελα να ρωτήσω τι είδους πραγματική δυνατότητα, τι είδους όγκους αφορούν. Ευχαριστώ κύριο Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα αν μου επιτρέψετε να μιλήσω όχι ως εκπρόσωπος της Πολωνίας, αλλά ως εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτη μου λοιπόν παρατήρηση. Τους συντονιστές τι τους χρειαζόμαστε εάν η μόνη τους δουλειά είναι να καταγράφουν μόνο τις συζητήσεις υπουργών. και πρωθυπουργών. Είναι δηλαδή περιτί εάν δεν μπορούν να ε, δώσουν ένα περιθώριο και επιλογές διαφορετικές από τα όσα θα πούν οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί και παρακαλώ να μην με ε, παρεξηγείτε, γιατί παρακολούθησα με προσοχή τη συζήτηση και για τις αγορές και για τις χώρες που πλήττει η κρίση και για το ότι η Πολωνία είναι η μόνη που παρουσιάζει θετική ανάπτυξη. Έγινε λόγος για αδυναμίες, έγινε λόγος για ελλείψεις, αλλά για ουσιαστική πρόοδο δεν άκουσα τίποτα. Στις 10 Νοεμβρίου έγινε μια συνάντηση των ε, Πρωθυπουργών ε, με τον Αντιπρόεδρο Κάλς και από ό,τι φαίνεται αυτή είναι η μόνη εξέλιξη των τελευταίων ε, εβδομάδων. Καλή εξέλιξη που θα τη χαρακτηρίσω, δηλαδή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε κάποια μετακίνηση της κυβέρνησης η οποία είναι πάντα αρνητική. Ένα πράγμα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορούμε να έχουμε ένα σημείο συνάντησης του, του ευρωπαϊκού με το ρωσικό δίκτυο. Υπάρχουν ε, εξελίξεις στη Λιθουανία, τη Λετωνία, ενώ στην Πολωνία δεν καταγράφεται πρόοδος. Έχουμε να κάνουμε με μια χρονική περίοδο 18 ετών που ξεκινήσαν τα σχέδια, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και τώρα πλέον χρειάζονται ήδη αναβάθμιση. Θεωρούμε λοιπόν εμείς σοσιαλιστές και δημοκράτες ότι δεν είναι επαρκής η πρόοδος, χρειάζεται να υλοποιούνται τα σχέδια. Είναι 15 χρόνια τώρα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Στην περίοδο αυτή η Λιθουανία και η Λετωνία παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη ε, της παρουσίας των διεθνών μεταφορέων, των διεθνών μεταφορών καλύτερα. 160.000 μεταφορείς εμφανίζονται μόνο στην Πολωνία στην περίοδο αυτή. Και γιατί, διότι επισκιάζεται και υπονομεύεται η συνδροδρομική μορφή των μεταφορών από τις λοιπές, από τα λοιπά είδη των μεταφορών. Θα θέλαμε λοιπόν συγκεκριμένα να μας πείτε ότι μόνοι σας δεν μπορείτε να τα καταφέρετε και πρέπει να βρείτε μια άλλη λύση. Ευχαριστώ, Ζήλα, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Τέλιτσκα ε, και να διαφωνήσω και με τον προλαλήσαντα συνάδελφο. Ε, ουσιαστικά με την σοσιαλδημοκρατική ομάδα διαφώνω για το θέμα αυτό. Για άλλα δεν μπορώ να κρίνω, αλλά σε ό,τι αφορά τον κύριο Τέλιτσκα και τη δουλειά που έχει κάνει για το Rail Baltica, πραγματικά το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, όταν πήγατε στη Ρίγα ήταν πριν την τελική δέσμευση της κυβέρνησης της Λετωνίας για να προχωρήσει με τη συγχρηματοδότηση και επηρεάσατε πάρα πολύ τα πράγματα, ασχίσατε πολιτική πίεση, ε, δημοσιοποιήσατε και μέσω των μέσων το πρόβλημα. Γι' αυτό και θα ήθελα να διαφωνήσω κάθετα με την ε, θέση των σοσιαλδημοκρατών σε ό,τι αφορά δηλαδή τη θέση των συντονιστών και δίκαια το συγκεκριμένο έργο. Τώρα, για αυτή τη μελέτη στο Intergroup της Βαλτικής ε, ε, υπάρχουν πολλοί που έχουν ακούσει τα σχετικά. Ε, το 2024 είναι το χρονοδιάγραμμα για αυτό το έργο. Θέλουμε να υπάρξει χρηματοδότηση και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκές πηγές και αν δει κανεί τι έγινε στι 10 Νοεμβρίου στο Ταλίν, ε, νομίζω ότι είναι θετικέ εξελίξει και θα συνεχιστούν. Έχω βέβαια και κάποιε αμφιβολίε, παρότι είμαι αισιόδοξο εν γέννη, αλλά οι αμφιβολίε μου υφίστανται και θα ήθελα να σχολιάσει ο κύριο ε, Τέλιτσκα. Ο Ντομπρόφσκη, ε, νυν και πρώην βέβαια Υπουργό, τέλο πάντων ανατυκλώνεται τα τελευταία χρόνια είπε ότι στηρίζουμε αυτό το ευρωπαϊκό project, αλλά θα πρέπει ε, η, με τη ρίγα να αλλάξει ε, η χάραξη, οπότε να είναι πιο ακριβό το project αυτό, όχι μόνο 3,3 δις, ή να βρεθούν περαιτέρω πόροι. Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο, ίσως δεν είναι και δυνατόν. Τι άποψη έχετε από αυτού. Και πραγματικά έχω κάποιες ε, αντιρρήσεις ό,τι αφορά αυτά, αυτές τις οικονομικές ομάδες συμφερόντων. Την προηγούμενη εβδομάδα δημόσια οι σιδηρόδρομοι της Λεπτανίας έχουν ε, ένα πρόγραμμα ηλεκτροδότησης ε, από Ανατολή προς Δύση δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν και το μεν και το δε έργο. Εσείς πώς βλέπετε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ήθελα να υπογραμμίσω ότι στις ε, εκθέσει αυτές που είδαμε βλέπουμε και αποφασιστική δέσμευση και σχετική πρόοδο την οποία οφείλουμε σε αυτή τη δέσμευση και τη στράτευση δική σας ε, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε και δεν μιλούμε για νέες ε, ε, διασυνδέσεις, μιλούμε για την διατήρηση της διασύγησης της, ε, των κρατών της Βαλτικής με την Ευρώπη ε, που περνούσαν πριν μέσω της Λευκορωσίας ενώ τώρα θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη διασύνδεση μέσω της Πολωνίας. Στην περίπτωση της περιοχής του Σουβάκη, ακόμα και μια μικρή ζώνη είναι μια καινούρια ε, γραμμή. Μπορεί να θεωρηθεί ως καινούρια γραμμή. 1,3 δισεκατομμύρια θέλουν οι Πολωνοί να αφιερώσουν στη μετάβαση, στην ε, μετακίνηση του φορτίου από το σιδηρόδρομο στις οδικές μεταφορές, ε, πράγμα το οποίο προσπαθήσαμε βεβαίως να παρεμποδίσουμε και ελπίζω να τα καταφέραμε. Ήθελα τα δικά σας σχόλια, πόσο, θα θα περάσει δηλαδή, και μετά βεβαίως η, το, το πλάτος της ε, τροχιάς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Ισπανία έχει κάνει την επιλογή της ε, πλατιάς τροχιάς. Στη συνέχεια, μετά τη Γαλλία, περνάμε στο ε, άλλο φάρδο, στο το κανονικό λεγόμενο ευρωπαϊκό φάρδος. Εδώ λοιπόν έχετε κάνει και εσείς την ίδια από ό,τι καταλαβαίνω επιλογή. Ωστόσο, έχετε μια νέα γραμμή, μια σύντομη διαδρομή καινούρια με την παραδοσιακή ευρωπαϊκή ε, συντηροτροχιά, ενώ από την άλλη πλευρά θέλετε να κάνετε επενδύσεις σε μεγάλου φάρδους σε φαρδιά σιδηροτροφιά. Δεν θα έχει κανένα νόημα αυτό γιατί θα μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και άρα θα ήταν καλό ε, να γίνει η επένδυση κατά τρόπο πιο ορθολογικό και που βέβαια θα επιτρέψει την κίνηση των τρένων ε, και από μεγαλύτερες αποστάσεις ώστε να ευνοηθεί και ο τουρισμός στις ώρες, αυτές τις περιοχές. Κόχλιτσεκ, τρία λεπτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε μετά από πολλά χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας, λοιπόν, κύριε Τέλισκα, και να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Στην ε, Τσεχία, όταν ε, φτιάχνουμε νέους διαδρόμους, 130 ε, χιλιόμετρα την ώρα είναι η ταχύτητα, ενώ στη Βαλτική είναι 120 χιλιόμετρα η ταχύτητα. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, και αυτό μου δημιουργεί έτσι κάποιες απορίες. Δεύτερο ερώτημα. Θα φροντίσετε αυτό το κομμάτι ε, να συνδεθεί με, με το πολωνικό κομμάτι, γιατί έχουμε κάποια προβλήματα με τις ε, τροχές και αν ε, δεν εξασφαλιστεί όλη η διασύνδεση αυτής εξ αρχής δεν έχει νόημα να προχωρήσουμε αυτό το έργο. Ξέρω ότι είστε ένας, αξιό, ένας ικανότατος διαπραγματευτής, άρα φαντάζομαι ότι έχετε προβεί σε απαραίτητες κινήσεις ήδη. Ευχαριστώ. Κύριε Τελίσκα, θέλετε να απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Έχω άλλη επιλογή κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω, λέει ο Πρόεδρος. Έτσι πάει το παιχνίδι, έτσι παίζεται. Μάλιστα. Ωραία κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας και θα απαντήσω με τη σειρά που μου ετέθησαν οι ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που είπατε το Rail Baltica, είναι σημαντικό έργο και για την Πολωνία. Είναι κάτι που ε, νιώθω κι εγώ ε, και το βλέπω όταν συνομιλώ με του ομολόγου μου στην ε, Πολωνία. Βέβαια ε, δεν είμαι αυτό ο οποίο θα έρχεται σε μια συνεδρίαση τη Επιτροπή για να λέει τι πέτυχε ή τι καταφέραμε γενικώ. Πρέπει να σα πω ότι ουσιαστικά τα κράτη-μέλη. Εγώ μπορώ να συντονίσω να ασκήσω κάποιες πιέσεις, να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Αυτό κάνουμε άλλωστε. Τώρα αν αυτό αρκεί ή όχι δεν θα το κρίνω εγώ. Δεν ήμουν εγώ αυτός ε, που πήγα στην Κομισιόν και είπα ότι θέλω να γίνω Ευρωπαϊκός συντονιστή, αλλά πράγματι για πάρα πολλά χρόνια, όπω είπατε, δεν έγινε καμία, ούτε μία εξέλιξη. Ακόμη και όταν το κόμμα σας ήταν στην κυβέρνηση στην Πολωνία. Φυσικά δεν μπορώ σε καμία περίπτωση τώρα να κάνω μια εξελιξη ακομη και οταν το κομμα σα ηταν στην κυβερνηση στην πολωνια φυσικα δεν μπορω σε καμια περιπτωση τωρα να κανω μια αξιολογηση του τι έγινε μέσα στην ε, πενταετία αυτή που ήταν ουσιαστικά μια προπαρασκευαστική φάση. Αυτό που βλέπω όμω είναι απτά αποτελέσματα και στην Πολωνία τα βλέπω και φαντάζομαι ότι υπάρχει πολιτική συνένεση επ' αυτού. Συμμετέχει και το κόμμα σας σε αυτή την πολιτική συνένεση και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέσα τα οποία επενδύονται. Ίσως την επόμενη φορά να δώσω πιο λεπτό, πολλές λεπτομέρειες στην αναφορά μου. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον θα τους ενδιαφέραν όλους οι τεχνικές λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι έχουμε επιτελέσει σημαντική πρόοδο στις χώρες αυτές. Αυτό είναι σαφές. Από τι μπορεί κανείς να το κρίνει, από τις συμφωνίες, από, την οικονομική, από τα οικονομικά μέσα. Πάντως, γύρω στο 2015 είναι σαφές ότι θα κυκλοφορούν σειρμοί τρένα τα οποία θα συνδέουν το Ταλίν με τη Βαρσοβία. Τώρα για το τι γίνεται στην Πολωνία. Θα έπρεπε ίσως να το είχα πει και το είπα και την περσίνη χρονιά και την προηγούμενη. Είπα ότι υπάρχουν αναβαθμίσεις. Γίνονται έργα αναβάθμιση ε, στην Πολωνία. Λυπούμε που δεν ε, σα έδωσα περισσότερες λεπτομέρειες από αυτού. Ό,τι αφορά τώρα την ε, διατροπικότητα και το σιδηρόδρομο, συμφωνώ μαζί σα. Δηλαδή πράγματι ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να ειδωθεί ως ε, φιλοπεριβαλλοντικός στρατηγικός βιώσιμος τρόπος μεταφορών. Στην Πολωνία και παράδειγμα στον κύριο Κράμερ, ναι μεν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, ε, η γραμμή δεν θα είναι ευθεία, ε, θα είναι λίγο υπάρχει μια κάποια παράκαμψη, αλλά υπάρχουν θεμητά προβλήματα περιβαλλοντικής φύσεως και αν χαθεί ένα τέταρτο ή τρία τέταρτα ε, μπορεί αυτή η καθυστέρηση να ανακτηθεί σε κάποιο άλλο κομμάτι του, του άξονα. Αν με ρωτήσετε αν έχω επιφυλάξει, εγώ δεν έχω, γιατί έργα γίνονται. Αυτό που θέλω να δω στην Πολωνία, και αν τα είπε και σωστά ο κύριος Ζήλε, πράγματι ε, ασκούμε ε, πολιτικές πιέσεις, γιατί θέλουμε να δούμε τα αποτέλεσμα στο στομότερο δυνατό αλλά δεν θα κρίνω εγώ. Επαναλαμβάνω. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι 15 χρόνια πέρασαν για να ξεκινήσει κάτι. Πολλές συμφωνίες, πολλά μνημόνια συμφώνησαν οι χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία, αλλά δεν έγινε τίποτα στην πράξη. Τώρα βλέπουμε να κινούνται τα πράγματα. Αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση. Τώρα, Σε ό,τι αφορά τι αμφιβολίε του κ. Ζήλε, δεν θέλω να βιαστώ, να διασκεδάσω τι ε, επιφυλάξεις γιατί είμαστε ακόμη στην αρχή. Αλλά κάτι έχουμε στα χέρια μας. Και αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι μια πάρα πολύ αναλυτική μελέτη σκοπιμότητας που δείχνει ότι είναι οικονομικά βιώσιμο το έργο. Ξέρουμε ότι είναι δαπανηρό. Αλλά τελικά μιλάμε για μια περίοδο μέχρι το 2024, ίσως και μέχρι το 2030. Εγώ, αν μου ζητήσετε τη γνώμη μου, θα πρότεινα το πιο αισιόδοξο σενάριο του 2024. Δύο δημοσιονομικές προοπτικές τουλάχιστον, αν λάβουμε υπόψη το 85% της χρηματοδότησης σε πραγματικούς όρους ή επιπτώσεις για τον πραγματικό προϋπολογισμό και σε καιρό ύφεσης, κατά την άποψή μου, είναι ανεκτές, γιατί είναι ένα στρατηγικό πρόγραμμα, στρατηγικό έργο. Δύο πολύ σημαντικά σχόλια που ακούστηκαν. Το ένα ήταν Ανατολή-Δύση. Πράγματι, αυτή η γραμμή είναι συμπληρωματική και θα ωφελήσει και, τη Rail, ε, και το Project Rail ε, Baltica. Αλλά για προφανείς οικονομικούς, ε, πολιτικούς και στρατηγικούς λόγους ο άξονας βορρά-νότου πρέπει να είναι ο σκελετός σπονδυλική στήλη. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό που βλέπουμε είναι πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευρά των επιχειρήσεων να εξετάσουν τι δυνατότητε σύγχρηματοδότηση κάποιων από τα κομμάτια του έργου που εκτελούμε. Μιλάμε για, αυτούς, για αυτό το κόμβο στο Κάουνα. και μία, αν θέλετε, ανόητη διελκυστίδα που υπάρχει μεταξύ δύο μήλων. Τελικά δεν έχουν συνειδητοποιήσει στην πραγματικότητα τι μπορεί να σημάνουν αυτά τα έργα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ότι θα προσελκύσουν επενδύσεις από το εξωτερικό. Επίσης μιλήσατε και για, τις, ε, για τα κονδύλια, για τα επιπλέον κονδύλια κύριε Ζήλε. Δεν μπορώ να σας πω ούτε πόσα ούτε αν και εφόσον. Εξετάζουμε ακόμη τις επιλογές αυτή τη φάση. Και εγώ μιλώ με την ιδιότητα του συντονιστή. Θα δω τον Αντιπρόεδρο στις αρχές Δεκεμβρίου και αυτό που θα ήθελα εν γέννη να συζητήσουμε είναι ότι εδώ μιλάμε για μια πραγματική στρατηγική ευκαιρία. Όχι μόνο για τις χώρες της Βαλτικής, εδώ μιλάμε για την ανταγωνιστικότητά μας απέναντι στις ε, χώρες Ανατολής. Δεν μιλάμε καν για την διασύνδεση. Λέμε, θα είναι ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές εταιρείε, θα ωφεληθούμε, θα έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη ή θα κερδίσει κάποιος άλλος. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και αν είχαμε περισσότερο χρόνο, θα μπορούσα ίσως λιγότερο διπλωματικά να σας δώσω μια πιο αναλυτική απάντηση. Τον κύριο Κράμερ, νομίζω ότι λίγο πολύ για το ΕΛΚ τα είπα, αλλά τώρα ε, σε ό,τι αφορά τη φάση, πόσο θα διαρκέσει, πρέπει να σας πω ότι περιμένουμε τη νέα πολωνική κυβέρνηση, ε, το σχηματισμό της νέας πολωνικής κυβέρνησης. Ε, θα πάμε σίγουρα στη Βαρσοβία και θα σχεδιάσουμε το έργο που πρέπει να γίνουμε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της επόμενης συμμετοχής προοπτικής, όχι των δύο, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Αλλά τις ε, λεπτομέρειες θα τις δούμε. Θα μας ε, πει και η μελέτη τα σχετικά. Εμείς πάντως θέλουμε να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί θα έχουν και ένα πολύ σωστό επιχείρημα οι χώρες της Βαλτική. Θα μας πούνε ότι εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Καταλαβαίνουμε ότι έχει λάβει μια θεμητή απόφαση και η Πολωνία. Θα πρέπει και αυτή να κάνει ε, αυτά που τις αναλογούν. Θα ζητηθεί αλληλεγγύη λοιπόν και ίσως να ασκήσουμε πράγματι και εμείς πιέσεις. Θα σας ενημερώσω, θα σας δώσω τα πιο συγκεκριμένα στοιχεία του σενάριου, της υπόθεσης ε, που θα επεξεργαστούμε όταν αυτά τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα αφού θα έχουμε συνομιλήσει με τις πολεμικές αρχές. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εν καιρό εκλογών και προεκλογικής εξαρτίας δεν ήταν τόσο εύκολο μέχρι τώρα. Επίσης μιλήσατε και για το νότιο τμήμα του διαδρόμου Βαλτικής Αδριατικής. Θα ξεκινήσουμε συνομιλίες με τις χώρες νοτίως της Πολωνίας άμεσα. Θα δούμε ποια είναι τα θέματα και σίγουρα μπορούμε φαντάζομαι να βασιστούμε και στη δική σας ε, βοήθεια. Είναι σημαντική η διάσταση η Βαλτικής Αδριατικής και μας δίνεται μια πραγματική ευκαιρία. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Κόχλιτσεκ, 130 χιλιόμετρα ε, στην Τσεχία, 120... Ναι, κοιτάξτε, πάντα πρέπει να γίνονται συμβιβασμοί με βάση συγκεκριμένες αναλύσεις και μελέτες. Αν πάρετε σήμερα ένα τρένο σε κάποια ε, σημεία στη Βαλτική, Μπορεί να πηγαίνουμε 30 χιλιόμετρα την ώρα, άρα και το 120 χιλιόμετρα είναι φιλόδοξο. Πάντως ο μέσος όρος μέσα ταχύτητα θα είναι 70 χιλιόμετρα. Επαναλαμβάνω, πιστέψτε με, θα είναι μεγάλη εξέλιξη αυτό. Όλα τα ερωτήματα του κύριου Κράμερ είναι θεμητά και λογικά, αλλά χρειαζόμαστε σίγουρα μια απλή γραμμή. Βλέπουμε τη συμπληρωματικότητα με την τρέχουσα. Πρέπει να ξεχρονιστεί η, η γραμμή. Το κόστος κατά την άποψή μας είναι εύλογο και σίγουρα θα αποφέρει κέρδος στο μέλλον. Και εγώ φαντάζομαι ότι θα εξοικονομηθούν και πόροι. Γιατί για τις ευρωματικές μεταφορές σε ένα βαθμό μπορεί να υπάρξει πλέον μεγαλύτερη ευελιξία με το Rail Baltica. Πάντω υπάρχουν σήμερα κάποιε προκλήσει. Πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε για το 2024. Τώρα δεν έχουμε εγγυήσει αν θα είναι έτοιμο το έργο το 2024 το 2030. Είναι μακρός ο χρονικός ορίζοντας, αλλά πρέπει να τον δούμε και από την πλευρά της εξοικονόμησης πόρων. Νομίζω ότι και τα δύο μπορούν να συνδυαστούν. Τώρα ποια θα είναι η γραμμή ακριβώς, σίγουρα αυτό είναι σημαντικό. Η χάραξη. Έχουμε δει την ένδειξη στο χάρτη, αλλά θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευθεία η γραμμή για να μειωθεί και το κόστος. Σαν διαφορετικά συνδεσιμότητα με την Πολωνία φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι απλά το εξετάζουμε, προσπαθούμε να το εξασφαλίσουμε. Άλλωστε, απλά και μόνο το ότι η Κομισιόν έλαβε την απόφαση να συνδυάσει το Rail Baltica, ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα διάδρομο Βαλτικής Αδριατικής, αυτή την κατεύθυνση δείχνει να ακολουθεί. Και άρα νομίζω διασκεδάζονται οι ανησυχίες σας. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε το λόγο. Κύριε Σάδα, θα σας δώσω το λόγο, αλλά να σας πω ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω. Δεν νομίζω ότι πηγαίνουμε ούτε με 130 χιλιόμετρα ούτε με 120. Ναι, με συγχωρείτε, δεν απάντησα μια από τι ερωτήσει για τον όγκο. Ναι, η Όγκη είναι όντω σημαντική. Πολύ ευχαριστώ να Ε, είναι, συγγνώμη, χαμηλή. Πολύ ευχαριστώ να σα δώσω κάποια στοιχεία. Αλλά αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι εφόσον δεν υπάρχουν υποδομέ, δεν μπορεί να κινηθεί ε, φορτίο. Η μελέτη ECOM που πολύ ευχαριστώ να σας δώσω δείχνει πιστεύω ποιοι μπορεί να είναι οι όγκοι στο μέλλον και δεν έχουν καμία σύγκριση με τους τωρινούς όγκους. Πολύ ευχαριστώ να σας δώσουμε τα στοιχεία. Okay. Thank you. Next, final one is priority project number six. This is the... Και προτεραιότητα παριθμών 6, Λιόν, Τριέστη, Κόπερ, Λουμπλιάνα, Βουδαπέστη, Ουκρανία, κύριε Μπρίνκχορστ. Και στο συγγνώμη σας καθυστέρησα λίγο. Ναι. ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω μερικά από τα σημαντικά θέματα που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Μόνο τα τελευταία, τις τελευταίες εξελίξεις. Θα σας αναφέρω. Μην, σταματάτε, μη συνεχίσετε. Θα ασχοληθώ εγώ με αυτά ε, στις κάρτες που ανεμίζουν στον αέρα. Πρόεδρε, αν ε, μιλούσαμε πριν από έξι μήνες, αντί για σήμερα, θα μπορούσα να είμαι πιο σαφής. Το σχέδιο προτεραιότητα 6 είναι πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία, όπω ξέρετε. Είναι η μόνη σιδηροδρομική γραμμή από Δύση προ Ανατολά και Τούμπαλιν, νοτίω των Άλπαιων. Άρα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ε, ρόλο. Μέχρι πριν από έξι μήνες λοιπόν ήμασταν σε ένα πεδίο μεγάλης αβεβαιότητας. Πλην όμως τον Ιούνιο του 2010 και με την συνδρομή του Αντιπροέδρου ε, Κάλλας ε, οι έξι χώρες Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, ε, Ουγγαρία υπέγραψαν το λεγόμενο μνημόνιο της Αραγώσα για να προσδιορίσουν τους όρους του σχεδίου αυτού. με τους όρους αυτούς και μην ξεχνάμε ότι μεγάλο κομμάτι του ε, επιχειρούμενου σχεδίου είναι, έχει ιστορική σημασία από τη Λιόν προς την Τριέστη δηλαδή. Ε, πιστεύουμε ότι και η ανάπτυξη του προς θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερα η Γαλλία και η Ιταλία έχουν διατυπώσει στρατηγικό συμφέρον για την υπόθεση αυτή θα θυμάστε ίσως τη συνθήκη του Τουρίνο του 2001 που αποτέλεσε και τη βάση τα τελευταία αυτά χρόνια πάνω στην οποία στηρίχθηκε, οικοδομήθηκε η πρόοδο στην υπόθεση αυτή. Για άλλα όμω θέματα που αφορούν πάντα την Ιταλία δεν σημειώθηκε η ίδια πρόοδος. Στο υπερμεθοριακό τμήμα στην περιοχή των Άλπιων, τη Γαλλία δηλαδή. Υπάρχει μια εξέλιξη με, ένα νέο, μια νέα σύραγγα 600 μέτρων και άλλες δύο στη Γαλλία και μία στην Ιταλία μικρότερες και επίσης μετά τις πολλές επιφυλάξεις ξεκίνησε η οικοδόμηση της σύραγγας το δε Αύγουστο εγκρίθηκε η φάση που αφορούσε την κοιλάδα Σούζα. Θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει η νέα κυβέρνηση. Συνεχίζω με την ε, συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας για τον περιορισμό του κόστους. Ξέρω ότι υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις και από εκεί. και ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα υπογραφεί και πριν δει το τέλος του έτους οριστική, στην οριστική της μορφή η συμφωνία. Η νέα Ιταλική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με το Σύμφωνο Σταθερότητας και έχει συμφωνήσει με το έχει βεβαιώσει το στρατηγικό συμφέρον, το στρατηγικό ενδιαφέρον του σχεδίου. Έτσι λοιπόν, αυτά όλα μπορούν να χαρακτηριστούν ως πρόσφατες εξελίξεις και θα ήθελα να ευχαριστώ από τη θέση αυτό κύριο Μάριο Βιράνο, ο οποίος με υπεράνθρωπες προσπάθειε, γιατί νομίζω ότι ε, δεν ήταν λιγότερο από 190 οι συνεδρίε των οποίων προείδρευσε τα τελευταία χρόνια, μα εξασφάλισε τη μέγιστη δυνατή συνένεση μεταξύ των πλευρών. Βέβαια, στους διαλόγους πάντα εκδηλώνονται πλειοψηφίε και μειοψηφίε. Είναι σαφές ότι με τη δουλειά του κύριου Βεράνο ε, έχει πιστεί έχουν πιστεί και οι τοπικοί πληθυσμοί. Η αποδοχή έχει πολύ μεγάλη σημασία, η περιβαλλοντική πτυχή έχει πολύ μεγάλη σημασία, η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πολύ μεγάλη σημασία και 10 από 24 δήμους σήμερα υποστηρίζουν τη σιδοδρομική αυτή γραμμή από τις τρεις κοινότητα που, κοινότητες που άμεσα επηρεάζονται από, την, ε, από, τα, από τα έργα, από την κατασκευή της γραμμής, οι δύο έχουν επίσης αποδεκθεί το σχέδιο. Ξέρετε ότι η ιστορική γραμμή που περνούσε από το Μονσενή είχε αρχικά αποτελέσει το, το αντικείμενο των συμφωνιών μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας και στο κομμάτι αυτό σύραγγα έχει, έχει ε, ανοίξει με τη νέα της μορφή, σε ορισμένα σημεία ακόμη με περιορισμένη ταχύτητα, αλλά προβλέπεται από 1η Ιανουαρίου του 2012 να λειτουργήσει πλήρως. Και η λεγόμενη προσέγγιση διαδρόμων που ανέφεραν και οι συνάδελφοι έχει πιστεύω ικανοποιητικά αξιοποιηθεί, γιατί στο ύψιστο επίπεδο εξασφαλίζεται συμφωνία για τις υποδομές που θα πρέπει να ε, αναπτυχθούν. Η πλήρη συνεργασία δείχνει επίσης και την πολιτική δέσμευση όλων των πλευρών και στη διαλειτουργικότητα που υπεγράμμισαν και οι συνάδελφοι γιατί ο σκοπό μα τελικά δεν είναι να έχουμε μόνο σιδηροδρομικέ τροχέ, αλλά διαλειτουργικότητα πάνω απ' όλα. Εδώ, Πρόεδρε, όλε οι εμπλεκόμενες πλευρέ, πιστεύω θα πρέπει να συμβάλλουν ε, και να ε, ε, συνεργαστούν κατά τρόπον ώστε να υπάρξει καλό συντονισμό, καλή συνεργασία για την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου στην, μέχρι την ολοκλήρωσή του. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Λίγα λόγια για την Ιταλία και τη Σλοβενία, Πρόεδρε. Η δυτική διάσταση δεν είναι πιο σημαντική από την ανατολική και δεν πρέπει να λησμονηθεί η ανατολική. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη φάση που αφορά την ανατολική διάσταση και η συνεργασία βεβαίως μπορεί να οδηγήσει σε μια ομάδα κοινών συμφερόντων για τις υποδομές που θα βεβαίω πιστεύω και με τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει με μετά τις εκλογές ε, τις επιλογές μας. Με την ελπίδα ότι στη γραμμή Λιόν Τωρίνο θα έχουμε την επιτυχία που αναμένουμε από τον Ιανουάριο και μετά μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα αποτελέσει αυτή η έμπνευση και για, την ανατολική, για το ανατολικό τμήμα της γραμμής. Επίσης για την Ουγγαρία θα θέλω να πω ότι στο πλαίσιο της ε, Ουγγρικής Προεδρίας και δι της ε, συνεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών το Φεβρουάριο συζητήσαμε το κομμάτι που αφορά την Ουγγαρία και την ανάγκη για περισσότερη διάρθρωτική συνεργασία μεταξύ Σλοβενίας και Ουγγαρίας ιδιαίτερως. Βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε κράτος προτιμάει να ορίζει με τη δική του εθνική κυριαρχία αυτές τις αρχές, αυτές τις επιλογές. Δεν είναι δεδομένη δηλαδή η ε, αποδοχή της διασυνοριακής συνεργασίας. Πριν όμω πιστεύω ότι μπορεί αυτή να αποδώσει καρπού μπορεί να έχει σημασία και αξία και ελπίζω να τη δούμε να αναπτύσσεται και μεταξύ Σλοβενία και Ουγγαρίας. Και ίσως από του χρόνο και μετά και χάρη στι αναμενόμενε επιτυχίες των λοιπών τμήματων τη γραμμή, πιστεύω να μπορούμε να χαιρετήσουμε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Σλοβενίας και της Ουγγαρίας. για το οικονομικό κομμάτι έχουμε ήδη προβλέψει σημαντικά ποσά. Και χάρη και στην προσωπική ανάμειξη του Επιτρόπου Κάλλα στα σχέδια αυτά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε περισσότερες ακόμη ε, σε μεγαλύτερη ακόμη πρικοδότηση του σχεδίου. Η ε, βελτίωση των υποδομών στην Ευρώπη, πρόεδρε, κλείνοντα, είναι πιστεύω μεγάλη επένδυση στο μέλλον τη Ευρώπη. Και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί με αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καντσάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συντονιστής μας, ε, Μπρίνκχορστ, ε, είναι αισιόδοξο και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Πιστεύει πραγματικά στην σημασία αυτού του διαδρόμου και μάχεται έτσι ώστε να επιτευχθεί το πέρας της οργάνωσης ενός τόσο δύσκολου περάσματος ανάμεσα στην Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ουγγαρία. Έκανα μια γενική, ε, ε, ε, κάνω μια γενική θεώρηση και μετά δύο ερωτήσεις για τον διάδρομο. και αυτές ε, οι γενικής φύσεως ε, παρατηρήσεις ε, ισχύουν και για τους άλλους συντονιστές. Όταν δουλεύετε για αυτούς τους διαδρόμους στα πλαίσια ενός, ενός συντονισμού πόσο βαραίνουν την, τις δυνατότητες σας οι τοπικές αρχές, οι πολιτικές αρχές, γιατί βεβαίως έχετε συγκεκριμένο ρόλο συντονιστικό και ε, βεβαίως ε, απέναντι σε δυσκολίες ε, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια μορφή εξουσίας και στον κόσμο που ζούμε πιστεύω ότι αυτές οι μορφές εξουσίας είναι υπερβολικά πολλές. Ε, ε, επομένως λέω ότι θα πρέπει να έχετε την δυνατότητα να μην είστε απλοί διευκολυντές αλλά συμμετέχοντες ουσιαστικοί στη λήψη απόφασης. Και εξού και η πρώτη μου ερώτηση πέρα από τις ε, γενικές δυσκολίες που απορρέουν το γεγονός ότι είναι διευρωπαϊκά τα δίκτυα αυτά ε, και, ότι είναι και διαλειτουργικά και που είναι φυσιολογικές δυσκολίες. Όμως ε, μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τις γραφειοκρατίες, μέσα από τις συνθήκες θα πρέπει να μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ήδη εμείς μιλάμε για τον προϋπολογισμό της, Ελλάδας, ε, της, συγγνώμη, της ε, Ευρώπης 2020, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για άλλα μη δημοσιονομικά στοιχεία. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι αυτά τα σχέδια, αυτός ο συντονισμός, αυτά τα προγράμματα να οδηγούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί έτσι επιβάλλουν οι καιροί και η κατάσταση που ζούμε τώρα είναι δραματική και ευαίσθητη. Κάνω λοιπόν έκκληση και στη δική σας καλή θέληση, αλλά κάνω έκκληση και στην πολιτική γενικότερα και σε εμά ακόμα τους ίδιους, έτσι ώστε ε, να έχετε δυνατότητες περισσότερες από αυτές που είχατε μέχρι τώρα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο διάδρομο, ε, αναφερθήκατε στο πέρασμα Βαλτισούζα και τις σχέσεις Ιταλίας-Γαλλίας. Ε, Ε, ωραία, ξεπεράστηκαν κάποια προβλήματα, αλλά έχουμε ε, βεβαίως και το τρία τη και αυτό είναι ε, δύσκολο. Εσείς βλέπετε η λύση να είναι, ε, δηλαδή μπορεί η οικοδόμηση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και για να ολοκληρώσω, η έκθεση του Επιτρόπου και άλλων Επιτρόπων μαρτυρεί την μεγάλη δέσμευση που έχουν αναλάβει οι Επίτροποι, αλλά δεν μπορούν, δεν έχουν εξουσίες έτσι ώστε να μπορούν να έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίπτωση. Επομένως ε, θα πρέπει να παίξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο σημαντικό ρόλο και λόγω των συνθήκων αλλά και βάση της διακυβέρνησης. Σαρικιάνη, Σαρικιάνη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με αυτά που μόλις είπε τώρα ο Καντσάνη βλέπω ας πούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Ιταλικό κομμάτι. Πού βρίσκονται κατά την άποψη του συντονιστή οι μεγαλύτερες δυσκολίες, οι σχέσεις με τους κρατικούς σιδηροδρόμους, με τις κυβερνητικές αρχές, τις δημοτικές αρχές. Γιατί οι διάδρομοι ενδιαφέρουν πολλές χώρες και επομένως θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκό μανδύα κατά κάποιο τρόπο και επομένως δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε υπερβολικά στις εθνικές ευαισθησίες και στην εθνική κυριαρχία. 26 υπογραφές από 11 διαφορετικούς οργανισμούς ε, χρειάζονται στην Ιταλία για ένα κομμάτι που το αντίστοιχό του στη Γαλλία χρειάζεται ας πούμε 5 αρχές και 2 υπογραφές. Εάν καταφέρουμε ε, αυτούς τους μεγάλους διαδρόμους να τους κάνουμε πραγματική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και ε, επομένως ε, να έχουν μια πραγματική υπερεθνική μορφή έτσι ώστε να ξεπερνούνται εύκολα τα, τα, εθνικά ή κρατικά προβλήματα, θα ήταν πολύ καλύτερα. Συγκεκριμένη ερώτηση. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και στο κομμάτι που φτάνει μέχρι τη Σλοβενία. Ελπίζω ότι και οι οικονομικές δυσκολίες ε, της ε, Σλοβενίας ε, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα σε αυτή την τροχιά. Και βεβαίως να πούμε ότι και η Ιταλία δεν είναι και ο καλύτερος μαθητής. Όμως υπάρχει ένα κομμάτι ε, Βενετίας ε, Τεργέστης ε, που δεν αναφέρεται πολύ συχνά. Οι αρχές, συνδεδοτικές αρχές θεωρούν ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό διότι δεν θεωρούν ότι είναι απαραίτητο. Έχετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες γι' αυτό γιατί πιστεύω ότι αν πραγματικά αυτή η πληροφορία είναι ορθή τότε δυναμητίζεται όλο το οικοδόμημα αυτού, αυτής της διαδρομής. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάτε για βελτίωση των υποδομών. Θα μπορούσα να σας... Ε, να συμφωνήσω μαζί σας ως προς τις υποδομές. Τα σχέδια όμως τα οποία δεν είναι αποδεκτά από τον πληθυσμό στις περιοχές αυτές θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Όπως είπε και ο συνάδελφο σας κύριος Μπάλλα, υπάρχουν πάντα εναλλακτικέ. Αυτό που γράψατε λοιπόν στην έκθεση για το παρατήριο και το κύριο Βιράνο, μπορώ να το δεχθώ μέχρι σε ένα σημείο. Ότι δηλαδή η έκθεση το 2010 προσδιορίζε προϋποθέσεις οι οποίες δεν ετηρήθησαν στο σύνολό τους. Εξού και το παρατηρητήριο και οι συζητήσεις προξένησαν τόσες πολλές ε, επικρίσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια επιλογή, μια γραμμική επιλογή ενδιαφέρουσα αλλά θα έπρεπε τη δέσμη αυτή είτε να την αναθεωρήσουμε είτε και να την εγκαταλείψουμε, διότι δεν αποτελεί τον πυρήνα βάσει το οποίο θα κρυθούν τα πάντα. Αυτή η, αυτό το, το σημείο συνάντησης δηλαδή δεν είναι το άπαν και θα μπορούσαν να βρεθούν διαφορετικές λύσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιμένουμε γιατί πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο και ό,τι και να λέει ο πληθυσμό, εμεί θα το επιβάλλουμε. Η Ιταλική κυβέρνηση χρειάστηκε να αποστείλει στρατιώτε ε, κατά χιλιάδε για να επιβάλλουν την τάξη. Αισθάνεται δηλαδή πολιορκημένο ο πολίτη στην ίδια του την πατρίδα. Και ναι, μεν πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι επίση υποστηρίζουν από πλευρά του το ε, σχέδιο, αλλά και αυτοί δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τι θέσει του. Εξού και θα ήθελα να πω, να ρωτήσω γιατί όταν γνωρίζουμε ότι είναι ένα σχέδιο τόσο διαφιλονικούμενο, γιατί δεν αναζητούμε εναλλακτικέ. Γιατί είναι απαραίτητο να επιμείνουμε σε κάτι το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό μόνο και μόνο γιατί είναι ευρωπαϊκό. Και ξέρετε επίσης ότι ο Ιταλικός Σιδηρόδρομος μόνο περισσότερες ε, ε, περισσότερα τρένα, περισσότερες διαδρομές, δηλαδή για μεταφορά επιβατών και μόνο από το Μιλάνο μέχρι την Νάπολη. Μόνο για τις επιβατικές μεταφορές. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες περιοχές και σε άλλες γραμμές. Το ξέρω πολύ καλά και από προσωπική μου εμπειρία και από τις ε, επιχειρήσεις που θα ήθελα να μεταφέρουν φορτίο σε αυτές τις γραμμές. Δεύτερον, θα γνωρίζετε πολύ καλά, φαντάζομαι, ότι για τις ε, εγκρίσεις χρειάζονται πολύ περισσότερα ε, δαπάνες από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και επίσης η Ιταλία ξέρω ότι δεν θα μπορούσε στο δική της κατάσταση την οικονομική να ανθέξει το βάρος όλων των επενδύσεων, αλλά δεν θα ήταν καλό τουλάχιστον να σχεδιάσει σωστά, δεν θα ήταν αυτό απαραίτητο για το για τις ευρωπαϊκές μεταφορές φορτίων. Ο κύριος Κόλτσικ παρακαλώ για τρία λεπτά μόνο. Ναι, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα. Πώς σκοπεύετε να πείστε ή πώς νομίζετε ότι μπορεί να πείσει η Ιταλική κυβέρνηση το κοινό ώστε να αποδεχθεί αυτό το σχέδιο. Και δεύτερον, Πώ θα συνδεθεί αυτός ο διάδρομος με τον άλλον πάει προς Βορρά, Τσεχία και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ, Ντάντε. Πρόεδρε. Ο κύριος Νταντάν, θα ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω κύριε Μπριγχόρστ για τη δουλειά σου όλη αυτή τη χρονιά. χάρη στι διαπραγματευτικέ σα ικανότητε, στι μεσολαβητικές σα ικανότητε, μπορέσατε να εξασφαλίσετε την, τις συνομιλίες και τη συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Και θα ήθελα αυτό, αυτού του γεγονότος να καταστώ εγώ προσωπικός μάρτυρας ενώπιον τη ομιλία. Ωστόσο, ε, τα καταφέρατε και τώρα πια πρέπει να περάσουμε και στην υλοποίηση. Είπατε σωστά κυρία Λεχτιμπέργκερ ότι υπάρχουν αμφισβητήσει, ότι υπάρχουν αντιδράσει. Αλλά δεν θα πρέπει και να μεγεθύνουμε την υπόθεση κατά τρόπον ε, ε, υπερβολικό. Εάν δούμε δηλαδή ότι αυτή η σύραγγα στην Ιταλική της την πλευρά έχει μετατραπεί σε ένα ε, σύμβολο αντίδρασης και αντίστασης στα ευρωπαϊκά σχέδια εν γέννη για ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι απλώς ο τοπικός πληθυσμός ο οποίος αντιδρά σε μία συγκεκριμένη σύραγγα που ενοχλεί συγκεκριμένα τρία χωριά. Όχι, αντιθέτω, ο πληθυσμό των χωρίων αυτών είναι πολύ θετικό ε, σε αυτή τη σύραγγα. Εδώ και τόσε ε, τι τελευταίε εβδομάδε έχουν τέτοια ατμοσφαιρική ρήπανση που έχουν ανεβάσει στο μέγιστο τον συναγερμό ρήπανση με υποχρεωτικό περιορισμό τη ταχύτητα στην περιοχή αυτή. Άρα σας διαβεβαιώ, οι τοπικοί πληθυσμοί είναι υπέρ της σύραγγας. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η σύραγγα όπως και όλες οι αντίστοιχες στις Άλπεις για τις ε, οδικές μεταφορές στην Ευρώπη. Και θέλω να ρωτήσω κύριε Μπρίνκχωστ, ξέρουμε ότι θα κοστίσει αυτό το έργο σημαντικά και πρέπει να συμβάλλουμε στην επιτυχία του από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του. Δεν θα πρέπει να έχει διευρυμένο λοιπόν ρόλο αυτό το, με χάρη, χάρη στην εντολή του ο διαπραγματευτής, ο, ο συντονιστής καλύτερα, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ουσιαστική υλοποίηση του σχεδίου, στην ε, από πρώτη στιγμή αξιοποίηση και αποδοτικότητα αυτού του έργου. Ευχαριστώ κύριο Σκράμερ, τελευταίες τρία λεπτά. Πρόεδρε. Θα σας πω το εξής κύριε συνάδελφε, κύριε η Ιταλία είναι σχεδόν στα όρια της πτώχευσης. Και βεβαίω είναι πολύ σημαντικά τα σχέδια. Υπάρχει όμως και μια ιεράρχηση. Ρότερταμ Γένοβα είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντικός ε, διάδρομος. Και σας διαβεβαιώ ότι εάν ε, διευρύνουμε την ε, εικόνα και κοιτάξουμε για στη Γερμανία τι γίνεται, ακόμα και στη, στο δρόμο Μόναχο-Σάλτσπουργκ δεν γίνεται τίποτα γιατί δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Στην, στην Ιταλία όμως φαίνεται δεν έχουν πρόβλημα να χρηματοδοτούν την Μπρεναβάζα ή την, ε, το, τη Λιόν Τωρίνο ή την γέφυρα στη Μεσίνη. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ιταλία είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν αυτά τα μεγάλα σχέδια και ξέρετε ότι η ιταλια ειναι σε θεση να χρηματοδοτησουν αυτα τα μεγαλα σχεδια και ξερετε οτι η χρηματοδοτηση άμα το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει ούτε το Κοινοβούλιο ούτε ο συντονιστής βεβαίως ούτε το Συμβούλιο καλά-καλά. Αποφασίσουν να χρηματοδοτήσουν παράλληλα διάφορα σχέδια χωρίς να μπορούν να τελειώσουν, αντί να επιλέξουν ένα και να το προωθήσουν. Πρέπει να γίνει μια ιεραρχική επιλογή και αν υπήρξε αυτή η ιεραρχική επιλογή, η προτεραιότητα δηλαδή, δεν θα ήταν η σύραγγα των Άλπιων η πρώτη επιλογή. Εκεί θα έπρεπε να κάνει διαφορετικές επιλογές η τελική κυβέρνηση. Εκεί θα έπρεπε και η νέα κυβέρνηση ακόμα της Ιταλίας ε, να προβεί σε διαφορετικές επιλογές. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπερλουσκόνη έχασε την ε, κυβέρνηση, έχασε τον έλεγχο της ε, κυβέρνησης, επειδή ακριβώς είχε φέρει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας τη χώρα. Και ίσως θα υπήρχε μία λύση η οποία θα πάρασε και από τα μεγάλα ε, φορτηγά των άνω των τρισιμιστών και θα επέτρεπε την ανάπτυξη οδών και διαδρόμων ε, πολύ πιο αποτελεσματικών. Ο Πρόεδρος. Δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο που θα υποστηρίζουμε την Ιταλία ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Κύριε Καντσιάν, 30 το πολύ να σας δίνω. Αλλά θα ήθελα να μείνουμε στην ουσία του θέματος, ε, όχι το κατά πόσον η Ιταλία ε, δεν ξέρω τι, τι συμβαίνει. Κύριε Καντσιάν. Ναι, ναι. Σας Κοιτάξτε, είναι ένα λανθασμένο σύστημα αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεν είναι ιταλικό το πρόβλημα ή ότι η Ιταλία ε, ε, προκάλεσε την αποτυχία. Μιλάμε για διάδρομο και αν έχουμε τέτοιου είδους πολιτικές και τέτοιου είδους θεωρήσεις, τότε δεν είναι διάδρομος αυτός από τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση, αρχίσαμε να δουλεύουμε για ένα διάδρομο. Δεν μπορούμε πλέον να γυρίσουμε πίσω. Δεν, δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα, γιατί διαφορετικά τότε ο διάδρομος δεν είναι διάδρομος, χάνει την ουσία του. Ας αφήσουμε, αφήσουμε λοιπόν την Ιταλία ήσυχη και ας δούμε ολόκληρη την Ευρώπη που βρίσκεται σε κρίση αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος. Ε, παιδιά, παιδιά. Παρακαλώ. Λίγη πειθαρχία, παρακαλώ. Η ε, κυρία Σαραγκιάννη θέλει τίποτα να πει. Όχι, έχουν υποθεί τα πάντα. Εντάξει, την Ιταλία την υπερασπιστήκαμε. Λοιπόν, ξέρουμε ποιε είναι οι απόψει του κυρίου Κράμερ ε, για την άνοιξη οπών μεταξύ Γαλλία και Ιταλίας. Τέλο πάντων, κύριε Μπρίγχορς, θα θέλατε να μας επαναφέρετε πλέον στο σχέδιο προτεραιότητας που αποτελεί αντικείμενό σας, κύριε Πρόεδρε. Τόσο πολύ ευχαριστήθηκα που θυμήθηκα και τότε που ήμουν Ευρωβουλευτής. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή γιατί δείχνει την πολυμορφία. Οι φίλοι μας μιλάνε για την Ιταλία, η Ιταλία αντιδρούν. Αυτά δείχνουν πάντως ότι είναι ενωμένη η Ευρώπη και πρέπει να είναι ακόμη πιο ενωμένοι λόγω και της κρίσης. Πρώτη απάντηση γενικού χαρακτήρα. Ο καθένας έχει ε, δικαίωμα να έχει τις απόψεις του. Ο κύριος Λιχτεμπέργκερ, ο κύριος Κράμερ, ο κύριος Κάντσιαν, ο κύριος Νταντά. Αυτές είναι οι πραγματικότητες όμως επιτόπου και με αυτές ε, πρέπει να ασχοληθούμε. Εγώ προσπαθώ να δεν ξέρω πώς να την πω αυτή την, ε, την παροιμία, αν κάποιος είναι κυβερνήτης, αν είναι πλοίαρχος σε ένα πλοίο, ο καπετάνιος είναι αυτός που έχει το πιδάλι στα χέρια του και όχι αυτός που κάθεται πιο πέρα. Λοιπόν, είναι σαν τον προπονητή τη εθνική αγγλία. Υπάρχουν εκατομμύρια που θα μπορούσαν να τα καταφέρουν καλύτερα από το Φάμπιο Καπέλο που αυτή τη στιγμή είναι προπονητή της Εθνική Αγγλία. Τέλο πάντων, εντάξει, δεν θέλω να φτάσουμε στο ποδόσφαιρο τώρα γιατί θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερο πάθο ε, και συναισθηματική φόρτιση και θέλω να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω για τα σχόλια και να πω ποιο, ποια σημασία έχει ο ρόλος του συντονιστή. Οι συνάδελφοί μου, ε, Μπάλας και Τέλης, έδωσαν ήδη κάποιες απαντήσεις. Εγώ να προσθέσω ένα καινούριο στοιχείο αν και εφόσον ανανεωθεί η συνθήκη του Τωρίνου, και ελπίζω να γίνει αυτό μέχρι τα τέλη του έτους, προβλέπει ότι η Κομισιόν, ε, λόγω του σημαντικού ρόλου που έχει στα οικονομικά, στη χρηματοδότηση, για πρώτη φορά σε ένα ευρωπαϊκό έργο θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η γαλλική κυβέρνηση, η γαλλική κυβέρνηση συμφώνησαν για πρώτη φορά να είναι στην, στο Διοικητικό Συμβούλιο η Κομισιόν. Είμαστε ο συνθητικό κρίκος. Δεν θα ψηφίσουμε κατά της μιας της άλλης κυβέρνηση. Ε. Ελπίζω να καταστεί σαφές ότι πέραν των γαλλικών ιταλικών συμφερόντων διακυβεύονται ευρωπαϊκά συμφέροντα. Η ευρωπαϊκή συνεργασία και η εθνική συνεργασία είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό μου έχει διδάξει εμπειρία μου τόσα χρόνια. Αλλά μετά από όλα αυτά τα χρόνια και με την εμπειρία μας, με τις ταλικές και Γαλλικές κυβερνήσεις. Και να πω για τις ταλικές κυβερνήσεις και της αριστεράς και της δεξιάς, έτσι. Και ο κύριος Πρόντι και ο κύριος Μπερλουσκόν, τώρα ο κύριος Μόντι, επιβεβαίωσε μάλιστα και ο ίδιος ο κύριος Μόντι ότι θέλει να ενταθεί σε αυτό το έργο ε, στο Σύμφωνο Σταθερότητας, βλέποντας ε, το στρατηγικό συμφέρον και μην κοιτώντας μόνο την ε, κρίση τη σημερινή. Αυτή άλλωστε ήταν η θέση μα πάντοτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία, νομίζω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια αναθεωρήθηκε το όλο έργο. Το είπα και στην κυρία Λίχτενμπεργκερ. Το έργο ήταν τελείω διαφορετικό στην αρχή. Η δημοκρατία υπάρχει, ισχύει, λειτουργεί. Η πλειοψηφία πρέπει κάποιε φορέ να σέβεται τι μειοψηφίε. Και βέβαια και οι μειοψηφίε πρέπει να σέβονται την πλειοψηφία. Έτσι γίνεται και στην πράξη. Η Ιταλία είναι ένα δημοκρατικό κράτο 14 κοινότητες ε, συμμετείχαν στις διαπραγματεύσει. 10 περιφέρειες είπαν ναι και από τις περιφέρειες οι δύο είπαν ναι. Στη χώρα μου πολύ λιγότερη ήταν η στήριξη του πληθυσμού σε ανάλογες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, δεν θα ε, αναφέρω τίποτε παραπάνω πάνω σε αυτό το θέμα. Φυσικά και πρέπει να έχει μεγαλύτερη ειδικό βάρος και η Κομισιόν και όταν θα ισχύσει η συμφωνία πλέον δεν θα έχουμε καμία αντιπαράθεση μεταξύ Γάλλων Ιταλών. Θα έχουμε ένα κοινό έργο που θα έχει κοινή διαχείριση και θα υπάρχει οικονομική συμμετοχή από την Κομισιόν πολύ σημαντική. Υπήρξε καθυστέρηση. Μάλλον δεν πρόκειται μέχρι το τέλος του 2013 να τα όλοι οι πόροι. Και η Κομισιόν ε, μάλλον είναι έτοιμη να παρατείνει για δύο χρόνια ακόμη την περίοδο. Για την κυρία Σαρακιάνη. Νομίζω ότι προσθέσατε ένα σημαντικό στοιχείο και κάνατε και ένα ερώτημα για την ε, Βενετία Τριέστη. Να σας πω ότι εγώ ήρθα σε επαφή και με τους ε, δύο περιφερειάρχες. Βέβαια αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με την εθνική διάσταση. Νομίζω τον Ιούνιο ή τον Μάιο συναντήθηκα μαζί τους και πραγματικά ανησυχούσαν ανησυχούσαν πραγματικά γιατί έλεγαν αν δεν γίνει τίποτε σε αυτό το μέρος ε, το να γίνει το επόμενο κομμάτι αν δεν υπάρχει η διασύνδεση μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού δεν έχει κανένα νόημα. Δεν ξέρω, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, είναι εθνικό το θέμα. Αλλά όπως ε, πάντοτε έτσι και τώρα μου δώσατε, με παρακινείτε και μου δίνετε ένα κίνητρο για να διερευνήσω την κατάσταση αλλά πρέπει να σας πω ότι στο κομμάτι ε, ε, Τριέστη Λιβάντζο έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος. Έχουμε εκλογές 4 Δεκεμβρίου, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ε, στη Σλοβενία, αλλά υπάρχει συνένεση να μπει ε, στον Όμιλο και τα τελευταίε στις τελευταίες εβδομάδες έχουμε κάποιες εξέλιξεις, αλλά λόγω των εκλογών δεν είχαμε κάποια τελική απόφαση. Θα με εξέπλητε πάντως αν η νέα κυβέρνηση, όποια σύνθεση και αν έχει, θα με εξέπλητε αν διαφοροποιεί το σε σχέση με αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα την κυρία Λίχτενμπέργκερ. Την απόψη μου την έδωσα, την είπα. Όπως είπα και πριν, ο καθένας μπορεί να έχει την απόψή του. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό για αυτήν την ιστορική γραμμή που επανασχεδιάζεται και το κατέστησα σαφές και στην εισαγωγή μου. 1η Ιανουαρίου έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ελπίζω στη μεγάλη αυτή χρονική περίοδο όσο θα ισχύει ακόμη η ιστορική γραμμή και μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί η νέα, ελπίζω να έχουμε και άλλες τέτοιες θετικές εξελίξεις για το περιβάλλον. Κόχλιτσεκ. Σε το συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι το ερώτημά σα. Μπορείτε να μου το επαναλάβετε. Το έγραψα, αλλά δεν το μπορώ να το διαβάσω. Πιστεύετε ότι η νέα κυβέρνηση θα έχει τρόπο και μέσα να πείσει τον πληθυσμό στην Βαλτισούσα και δεύτερο ερώτημα η διασύνδεση αυτού του διαδρόμου με το διάδρομο που περνά από την Τσεχία, την Πολωνία, Σλοβενία. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ζητώ συγγνώμη, ο κύριο Μπρίνκχορστ, για τον πρώτο. Είπα και πριν από δύο-τρία λεπτά. Επειδή θέλω να είμαι βέβαιο ότι η κυβέρνηση Μόντι θα πάρει την ίδια θέση, το έλεγξα το σημείο αυτό. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι στρατηγικό ε, το έργο αυτό και πρέπει να συνεχιστεί. Δεύτερον, πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι τίθεται για πρώτη φορά. Φυσικά, είναι προφανές ότι αν η γραμμή μεταξύ Σλοβενίας-Ουγγαρίας περάσει, φτάσει στην ε, Ουκρανική μεθόριο, κάποια κομμάτια της δεν λειτουργούν, ούτε καν ηλεκτροδότηση δεν υπάρχει σε μερικά και άρα αυτό συνιστά ένα σημαντικό περιορισμό. Σίγουρα ε, επηρεάζεται η όλη διασύνδεση προς βοράν. Τώρα έχουμε επιλέξει την προσέγγιση του διαδρόμου και η Κομισιόν το στηρίζει, το στηρίζει στεναρά. Ελπίζω λοιπόν να το στηρίξουν το έργο αυτό και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και θα ήταν χρήσιμο να γίνει ένας πολύ πιο εντατικός διάλογος μεταξύ, για τους διαδρόμους ε, Βορρά, Νότου και Δύσης Ανατολής. Η Βουδαπέστη είναι πάρα πολύ ε, σημαντικός κόμπος και παραδοσιακά και ιστορικά στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. Άρα θα έχει προσθεμένη αξία για το έργο. Για τον κύριο Νταντέ εν τέλει θέλω να τον ευχαριστήσω για την υποστήριξή του ως προς το σχέδιο αυτό. Ήταν υποδεγματική κατά το παρελθόν η γαλλική κυβέρνηση. Έχουμε αυτά τα διερευνητικέ αυτές σύραγγες που ολοκληρώνονται και υπήρξε και ανακούφιση από τη γαλλική πλευρά. Πλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις, άρα μπορεί να ξεκινήσει το έργο και να υλοποιηθεί. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Brinkhorst, Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις, ε, Μπάλα, Στελίτσκα, Brinkhorst για τις παρουσιάσεις που έκαναν για αυτά τα έργα προτεραιότητας και για τις απαντήσεις που έδωσαν και για την τροφή που έδωσαν για συζήτηση και για τη διαφωνία μεταξύ Επιτροπής ε, Μεταφορών Τουρισμού. Δεν είναι και πολλοί αυτοί που μπορούν να το καταφέρουν, αλλά κάνει καλό στην ψυχή έτσι και ένα τσακωμός. Εμείς στην Επιτροπή Μεταφορών ε, θέλουμε τα αποτελέσματα και γι' αυτό συνεργαζόμαστε και θέλουμε να συνεργαστούμε. Καταλαβούμε τις δυσκολίες που έχετε να αντιμετωπίσετε με κάποια από τα κράτη-μέλη. Και εμάς το ίδιο μας ενοχλεί και μας απογοητεύει κάποιες φορές η κατάσταση με κάποια κράτη-μέλη. Θα ακούσουμε και κάποιους από τους συναδέλφους σας αύριο, που φαντάζομαι θα επαναλάβουν ε, τα ίδια λόγια απογοήτευσης, αλλά εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε και ελπίζουμε να έχουμε και να πετύχουμε. Κρατάμε την μπάλα στα πόδια μας, κάνουμε και κάμια τρίπλα και θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Λοιπόν, ευχαριστώ να πω στους συναδέλφους ότι θα δούμε τώρα τα διάφορα, γιατί αύριο δεν θα είμαι εδώ. Πείτε το, ίσο πάστε για πάντα. Έχετε κάτι στα διάφορα. Όχι, άρα λίγη σημερινή συνεδρίαση. Και σας ε, υπενθυμίζω αύριο στις 9 ε, επαναλαμβάνονται οι εργασίες μας με τον ε, Πατ Κόκ, την Κάρλα Πέις, με ανταλλαγή απόψεων και με τον Επίτροπο Κάλλας στις 12 το μεσημέρι και στις 11 ο αγαπητός συνάδελφος αντιπρόεδρος Ρικέ θα προεδεύσει από τις 11 και μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.